Okay, colleagues, can I bring the meeting to order before we go into the hearing on the airports package at half past three? We. Ο πρόεδρος. Ήρθε η ώρα και έχουμε στις 3.30 την έκθεση του κ. Πάνιου ε, όσον αφορά κάποια οχήματα. βλέπω τον κύριο εισηγητή, κύριο Πανιόλ, και έχει το λόγο. Συνάδελφοι, λέει ο κύριος Παρνιό, έχουμε αυτή την, το, το, σχέδιο πρόταση κανονισμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, όσον αφορά αυτά τα μηχανοκίνητα οχήματα. Λεωφορεία, ε, ημιφορτηγά ε, και βαρέα φορτηγά και έχουμε τις σχετικές εκπομπές που κανονίζονται, ρυθμίζονται από κάποια οδηγία. 70-57 και θέλει να επικαιροποιήσει αυτό το νομικό πλαίσιο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βασική στόχη είναι πρώτα-πρώτα η απλούστευση της νομικής ρύθμισης, του νομικού πλαισίου και έτσι με αυτή την οδηγία να να, να έναν κανονισμό παλαιότερο, επίσης να έχουν μια καινούργια μέθοδο για τις ε, δοκιμές σε σχέση με τα όσα από το 2007 εθέσπισε ο ΟΗΕ και να πάμε σε εκπομπές κάτω από 2 δεσιμπέλ σε επίπεδο θορύβου σε σχέση με τις προηγούμενες οδηγίες και θα, αυτό θα ισχύσει για κάποια περίοδο κοιμής τριών ετών και, και τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιοποίησε την ε, μελέτη των επιπτώσεων και προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γίνει μια προοδευτική, ε, προοδευτικός υπολογισμός αυτών ε, και να έχουμε 4 δεσιμπέλ πραγματικά 5 χρόνια μετά τη θέση ισχύ του κανονισμού. Σε δύο χρόνους πρώτα πρώτα κάτω από τα δύο για το 2014 και σε μια δεύτερη επιτροπή κάτω από τα δύο με στόχο το 2017. Τα δε επίπεδα των ηχητικών εκπομπών ανά όχημα να μην ξεπερνάνε τα 68 τελικά δεσιμπέλ για τα βαρέα οχήματα. Τώρα 3 στα 5 χρόνια 3 δεσιμπέλ μόλις ε, τεθεί σε εφαρμογή το η νομοθεσία και κατόπιν έχουμε το 2014 μείωση κατά 1 και 2 με στόχο το 2017. Οπότε να μην ξεπερνάει τα 78 τελικά. Ε, επίσης να έχουμε ένα ελάχιστο επίπεδο θορύβου για τα ηλεκτρικά οχήματα και τα υβριδικά. Και έτσι να εξασφαλιστεί ότι μόνο όσα κρίνονται επαρκή να χρησιμοποιούνται και να παραμείνει να παραμείνουν και αυτές οι ρυθμίσεις κατασκευής ενδοτικού δικαίου για τους κατασκευαστές. Έχουμε τώρα αυτά τι τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχουν υποβληθεί σε αρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου για να δούμε κατά πόσο είναι εφικτή η στόχη. Έχουμε κάποιες ε, προτάσεις τροποποίησης αυτού του κανονισμού που αφορούν τα εξής σημεία. Πρώτα-πρώτα, πρώτη τροποποίηση, προσθήκη των οχημάτων με δύο ή τρεις τροχούς και σε σχέση με τον επόμενο κανονισμό δεν έχουμε ε, καμία ρύθμιση για τα δίτροφα και τρίτροφα. οπότε υπάρχει εδώ νομοθετικό κενό και γι' αυτό θα πρέπει να πούμε ότι χρειάζεται να πάνε η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ούτω ώστε έτσι να καλυφθούν αυτά τα δίτροφα και τα τρίτροφα. Η δεύτερη τροπολογία ε, καινούριε οριακέ τιμές όσον αφορά τα βαρέα οχήματα και θα πρέπει επίσης να δούμε κατά πόσον για τα ελαφρά οχήματα, να, συμφωνώ για τα 4 δεσιμπέλ για αυτά τα 7 χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ του οργανισμού. Οπότε αυτή η μείωση θα γίνει σε δύο φάσεις. Πρώτος στόχος κάτω από τα 2 δεσιμπέλ το 2014. Στη συνέχεια δεύτερη μείωση να κατέβουμε άλλα 2 ε, το 2019 και για τα βαρέα οχήματα να συμφωνήσουμε προτείνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τρίτη τροπολογία να έχουμε για τα ηλεκτρικά και τα υβριδικά μια ρύθμιση και γιατί έχουμε ε, στις, στις πόλεις ε, μπλέκονται σε ατυχήματα δύο-τρεις φορές δυστυχώς. Και αυτό γιατί επειδή δεν κάνουν θόρυβο, οι τυφλοί και οι κουφοί δεν τα βλέπουν και δεν τα ακούνε. Και οπότε θα πρέπει να υπάρχει τελικά κάτι σαν κλάξον, τόσο κάτι να προειδοποιεί και αυτό να είναι υποχρεωτική η ρύθμιση και να μην είναι ενδοτική η ρύθμιση αυτή όπως το, το, το, το, το θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίση, όσον η δική μα επιτροπή, να έχουμε και κάποιε επιπλέον τροπολογίε για να τροποθεί το κείμενο. Να δούμε με ποια στοιχεία μπορούμε να σταματήσουμε την ηχορύπανση. Ε, σε σχέση με τα λάστιχα, τα χήματα και επίσης καθές. Και έτσι θα πρέπει να δούμε πώς θα υπάρχει όσον αφορά την πώληση, θα υπάρχει ε, διαφάνεια όσον αφορά τους καταναλωτές καθές. Και επίσης θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα ανώτατα όρια σε σχέση με τα διαφορετικά είδη οχήματος πέραν των 90 δεσιμπέλ. Ακριβώς όπως ε, προείπα, μέσα στις 15 του μηνός έχετε το μεσημέρι, ούτως ώστε να καταθέσετε τροπολογίες. Και στη συνέχεια, στην Επιτροπή μας ε, στις 18 Ιουνίου θα το συζητήσουμε και θεωρητικά την επόμενη μέρα, δηλαδή στις 19 Ιουνίου θα γίνει η ψήφιση στην Επιτροπή μας. Αυτά, πρόεδρε και συνάδελφοι, αυτά που ήθελα να σας εξηγήσω όσον αφορά την ονομοδότησή μου. Σας ευχαριστούμε πολύ, λέει ο κύριος ε, Σίμψον. Και τώρα έχουμε τους ε, σκιώδους ηγετάς. Όμως, συνάδελφοι, πρέπει στις 3.30, όπως προβλέπετε, να αρχίσουμε την ακρόαση. Όμως, πρώτα-πρώτα, σκιώδους ηγετές. Κύριος Κόζα για την... Η κυρία Κόζα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα πρώτα-πρώτα, λέει ο κύριος Γκρός, να συγχαρώ τον εισηγητή. Άρεστη η δουλειά του ε, και ήταν η παρθενική του έκθεση και συμφωνώ με τις τροπολογίες του. Δεν ε, μπορέσαμε να συνοηθούμε, να έρθουμε σε επαφή νωρίτερα, όμως είμαι βέβαιος ότι στη συνέχεια θα συνεργαστούμε όπως πρέπει. Είναι πάρα πολύ σημαντική η έκθεση και το θέμα αυτό. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε απλούστευση της ρύθμισης και έτσι θα ενισχυθεί η υπόθεση της προστασίας κατά ε, του θορύβου. Ε, ήμουν εις να μιλήσω με διάφορους από τους εμπλεκόμενους από την σχετική βιομηχανία και τα συμπεράσματά μου από τις επαφές μου ήταν τα εξής. Να σας πω τι έμαθα από αυτούς. Πρώτα πρώτα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει κάποιο σύστημα δικτύωσης. Να είναι απλό και γρήγορο. Άρα να εξετάσουμε έτσι κάποια θέματα τα οποία δεν έχουν ξεκαθαριστεί. Δηλαδή η ποιότητα των ελαστικών των οχημάτων. Γιατί και τα ελαστικά ανάλογα με το υλικό από το οποίο προέρχονται δημιουργούν και αυτά θόρυβο. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξεταστεί ό,τι ήδη ισχύει. Δηλαδή, τα οχήματα που ήδη έχουν παραχθεί. Θα πρέπει οι μετρήσεις να γίνουν ακριβέστερες. Αν κάνει εξετάσει τι ωριακέ τιμέ έχουν δεσπιστεί, τότε θα διαπιστώσει ότι αυτές οι ωριακέ τιμέ είναι αποδεκτέ από όλους τους ε, εμπλεκομενου ομως Όμως έχουμε δύο θέματα πάρα πολύ επίμαχα. Πρώτα-πρώτα για τα υβριδικά. Διότι η πρώτε Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποσκοπεί ή στο να υπάρχει ένα καθορισμένο όριο ή επίπεδο θορύβου. Αυτό προσέχει ενδιαφέρον ότι δηλαδή τα συνήθεια οχήματα εάν περνούν από τεχνικό έλεγχο να είναι λιγότερο θορυβόδη από τα υβριδικά. Άρα να είναι αρκετά ευέλικτε οι τελικέ ρυθμίσει. Κάτι άλλο τώρα. Δεν προκύπτει την έκθεση ξεκάθαρα το θέμα του, των ορίων ταχύτητο. Όσο πιο γρήγορα οδηγεί κανεί, πιο πολύ θόρυβο δημιουργεί. Θα πρέπει βεβαίως να λάβουμε υπόψη και ε, τα θέματα που αφορούν τους τυφλούς. Θα πρέπει δηλαδή να είναι υποχρεωτική ρύθμιση που αφορά το επίπεδο θορύβου που, που, που, δημιουργείται. Από την άλλη μεριά βέβαια υπάρχει το, το θέμα της προειδοποίησης των τυφλών και, και άλλων αναπήρων όπως των κοφών. Ή τόσο όσων έχουν δυσκολίες στην ακοή γιατί και εκείνοι θα πρέπει να μπορούν να καταλάβουν ότι πλησιάζει ένα όχημα το οποίο αποτελεί κίνδυνο. Ελπίζω ότι με συμβασικές τροπολογίες όλα αυτά θα τα ρυθμίσουμε. Σας ευχαριστούμε. Τώρα η σειρά των φιλελευθέρων. Κύριε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Λέει η κυρία Σαββισάρ. Συνάδελφοι. Το επίπεδο εκμεμπημένου θορύβου από τα οχήματα είναι ένα θέμα σημαντικό και με τη ρύθμισή μας θα πρέπει να καλύψουμε όλους τους εμπλεκομένους, να δούμε τι θα γίνει και με την ε, ρήπανση του περιβάλλοντος. Ο κόσμος φυσικά θέλει ε, μια καθαρή ατμόσφαιρα και επομένως εκεί υπάρχει κόκκινη γραμμή όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της ρύθμισης. Τώρα όσον αφορά το σχέδιο κειμένου δυστυχώς ο εισηγητής δεν πρόσεξε κατά τη γνώμη μου ε, τις θέσεις τις δικές μας, των φιλελευθέρων. Και δεν δε, ούτε καν συναντήθηκε με διάφορους από τους σκιώδεις εισηγητές. Φαίνεται σημαντικό να έρθουμε σε επαφή μαζί του, διότι ο περιορισμός του επίπεδου του εκπαιδευμένου θορύβου ε, είναι κάτι το οποίο καίει και τους λομπίστες και, τους, ε, και τις Όσον αφορά τώρα τα βαρέα οχήματα, είναι θέμα κατάταξης χαρακτηρισμού, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας προτείνει δύο κατηγορίες. Πρώτα-πρώτα, ε, με ισχύ κινητήρος κάτω από τα 150 κιλοβάτ και ε, τα, τα υπόλοιπα οχήματα είναι η δεύτερη κατηγορία κάτω από το όριο. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε τρεις κατηγορίες. 180 κιλοβάτ και 250 και με, ε, κάτω από 180, ε, μετά 180-250 και τα υπόλοιπα τρίτη κατηγορία πάνω από 250. Από την άλλη μεριά, το μέγεθος του οχήματος δεν συνδέεται άμεσα με τις δυνατότητες της, ε, της μηχανής, του κινητήρα. Και αναφέρομαι τώρα ή στα λεωφορεία. Τέλος πάντων, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής και ισχύω του, του, του, της ρύθμισης. Θα πρέπει να δούμε αν η βιομηχανία μπορεί να ανταποκριθεί, αν μπορούν να παράξουν αυτά τα αυτοκίνητα τα οποία θέλουμε. Δηλαδή, αν θέλει κανένα σήμερα ένα όχημα καινούριο, ε, δεν γίνεται. Πρέπει να περιμένει 12 μήνε, ένα χρόνο. Μπορεί δηλαδή να, προσαρμοστεί η βιομηχανία αυτό που ζητούμε και, και σε, σε χρόνια ε, από την άλλη μεριά δεν είχε αιτιολογήσει επαρκώ ο εισηγητή τι προτάσει του. Γιατί νομίζει ε, ότι χρειάζονται άλλε ρυθμίσει για τα γεωταχή, για, για τις, μικρότερου κινητήρε, Γιατί μα λέει 1900 κυβικά εκατοστά ω επιπλέον όριο στο μέγεθο του κινητήρα. Νομίζω ότι το μοναδιαίο κόστο είναι χαμηλότερο για τα γεωταχή παρά για τα άλλα οχήματα, για τα λεωφορεία α πούμε Υποτελεί θα σε επαφή με τους εμπλεκόμενους. Όμως, αυτοί είπαν αντίθετα. Ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν συντονίστηκε μαζί τους. Ούτε θα σε επαφή με τον φορέα των Ευρωπαίων αυτοκινητοβιομηχάνων. Επίσης θα πρέπει εκτός από τη μόλυνση και τη ρήπανση να προσέχουμε και την αποτελεσματικότητα των μεταφορών να μην προσέχουμε μόνο του κινητήρε, αλλά και το σχεδιασμό του αυτοκινήτου, το design και τα ελαστικά. Να είμαστε δίκαιοι με τον κύριο Πανιόλ και του συμπατριώτες του. Σχετικά με το αν ήρθαν σε επαφή με του άλλου εμπλεκόμενου, είμαι σίγουρο ότι θα το κάνει τι αμέσως επόμενες εβδομάδες ο κύριο Πανιόλ. Από την άλλη μεριά, τις τελευταίες δύο εβδομάδες οι Γάλλοι συνάδελφοι, όπως ξέρετε, είχαν άλλα θέματα. Ήταν οι εκλογέ τέλο πάντων. Παρακάτω, Τέιλορ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το κείμενο του. Σήμερα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, η χορύπανση η έρχεται δεύτερη μετά την ατμοσφαιρική ρήπανση όσον αφορά τις συνέπειες. 210 εκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εκτεθειμένοι εις ε, επιβλαβή επίπεδα θορύβου. Επίσης, με εξέλιξε το ότι λέει, έχουμε 50.000 πρόωρους θανάτους σε σχέση με το, το θόρυβο από, από την κυκλοφορία. Και επίσης έχουμε πάρα πολλέ περιπτώσεις καρδιαγγειακών παθήσεων. Γι' αυτό σας λέω, μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε αποτελεσματικά μέτρα, ούτως ώστε να μειώνονται τα επίπεδα θορύβου των ε, οχημάτων με κινητήρα ή στου Ευρωπαϊκού δρόμους. Δυστυχώ. οι προτάσει τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεωρώ ότι είναι ανεπαρκείς, ούτω ώστε να ε, οδηγήσουν σε προστασία της υγείας, μείωση του κόστους μέσω της μείωσης του εκπαιμπωμένου θορύβου από τα οχήματα. Οπότε για αυτό το λόγο και οι πράσινοι πρόκειται να υποβάλουν τροπολογίες για την ε, ε, έκθεση του κυρίου Παρνιό σε σχέση με τις διατάξεις 10 και 13. Επίσης είμαστε και σε διαφωνία και με άλλους προλαλήσαντες. Επίσης δεν θέλουμε να καθυστερήσει η θέση ισχύ του κανονισμού, γιατί έτσι θεωρούμε ότι θα αποδυναμωθεί το επίπεδο ρύθμισης των υπομένων δεσιμπέλ. Με τις τροπολογίες μας θα εξασφαλίσουμε το ότι παρεκκλήσεις θα βρίσκονται στα, στα τρία χρόνια μόνο μετά την θέση σε ισχύ. Και επίση κάποιε ρυθμίσει θέλουν να μείνουν για τα τετράτροχα και όχι για τα δίτροχα. Για άλλη μια φορά επίση, προβληματιζόμαστε όσον αφορά το πόσο ε, παραμελείται το περιβάλλον, γιατί σας ξαναλέω ότι δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο, τίποτα που να σκοτώνει περισσότερο από τον θόρυβο που εκπέμπουν τα αυτοκίνητα, ε, γενικά ο θόρυβο, παρά μόνο η ατμοσφαιρική μόλυνση, ρήπανση, φώστερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και να ευχαριστήσουμε και τον εισηγητή, λέει η κυρία Φώστερ. Έχετε δίκιο. Το πιο σπουδαίο τώρα είναι να κάτσουμε και να τα συζητήσουμε. το ότι δημιουργώντα την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι δεν καταλαβαίνω από πού ξετρύπωσαν όλα αυτά τα στοιχεία για την μείωση. Καλά λέμε για 30 συμπέλη, ξέρω εγώ τι λέμε, αλλά αυτό το οποίο θα πρέπει να λάβει κανεί υπόψη του είναι το πώ θα πετύχει αυτό που θέλει. Δεν λαμβάνουν υπόψη του ένα χρονικό πλαίσιο λογικό. Τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει ένα μηχανικό. Θέλουμε να μειώσουμε το θερμό του κινητήρα. Αλλά προσοχή γιατί πάνε σημείο και πέρα αναβαίνει η κατανάλωση του καυσίμου. Άρα το ένα μην ακυρώνει το άλλο. Αυτό το οποίο εμείς πρέπει να κάνουμε είναι μαζί με το θόρυβο να δούμε τις υπόλοιπες συνέπειες. Και επίση το πιο σωστό είναι οι προτάσει της Κομισιόν να είναι ρεαλιστικές που με αυτό το χρονισμό που, που λαμβάνει υπόψη η Κομισιόν δεν τις κάνει ρεαλιστικές. Σύμφωνοι. Έχω στην εκλογική μου περιφέρεια αυτοκινητοβιομηχανίες δεν σα το κρύβω. Και έχω μιλήσει μαζί του όμω για να μάθω τι είναι εφικτό και τι δεν είναι. Η Κομισιόν όμω μίλησε με κανέναν. Επίση, μου φαίνεται πάρα πολύ προσβλητικό όταν στην πρότασή του περιλαμβάνουν κάποια στοιχεία που λένε για το τι προτείνει η μελέτη επιπτώσεων όσον αφορά τα ωφέλη της υγεία και λέγεται για 117 δις μέχρι το 2030. Πού τα βρήκαν αυτά. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε μια συζήτηση χωρίς να, να, να, τρομάζουμε τον κόσμο. Εδώ μας φαίνονται σαν να είμαστε νηπιαγωγείο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρουμε για όλα αυτά τα θέματα ότι υπάρχουν επιπτώσεις, αλλά δεν να μας πετάνε κάποια τέτοια στοιχεία τα οποία κύριος είδα που προήλθαν. Ναι, να μειωθεί ο θόρυβος. Όχι, δεν σα τα λέω αυτά για, κομματικό συμφέρον, αλλά δεν θέλω και να κλείσουν και τα εργοστάσια που είναι στην περιφέρειά μα. Προσοχή, γιατί πρόκειται για ένα τεράστιο κλάδο, πολύ σημαντικό σε απασχόληση, πολύ σημαντικό για την έρευνα κλπ. κλπ. Οπότε γι' αυτό και ελπίζω ότι η Επιτροπή Μεταφορών να είναι πραγματική Επιτροπή Μεταφορών και τελικά να καταλήξουμε σε κάποια πρόταση λογική. Πώς το με κύριε Φώστερ, λέει ο πρόεδρος. Λαγκράν. Ο κύριος Λαγκράνος που εκπροσωπεί την Κομισιόν. Δύο λεπτά δεν στο λένε να σας ζωρίσω, αλλά έχουμε κοντζά μακρόες στη συνέχεια, γι' αυτό σας το είπα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Α, αγαπητοί κύριοι βουλευτές, που να ευχαριστήσουν πρώτα-πρώτα την Επιτροπή σας γιατί μας δίνει την ευκαιρία να σας πούμε την άποψή μας για το σχέδιο της γνωμοδότησης. Ναι, ναι, πρόεδρε, προσπαθώ να είμαι σύντομος. και το πρώτο το οποίο θέλω να σας πω είναι το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, όπως το είπε ο εισηγητής. Ο κανονισμός μας δεν θα καλύψει δίτροχα ή τρίτροχα. Και για αυτό γίνεται διότι έχουμε άλλο νομοθέτημα που καλύπτει δίτροχα και τρίτροχα. Πρόκειται για κανονισμό πλαίσιο που τώρα βρίσκεστε στη διαδικασία εξέτασή του για τα δίτροχα και τρίτροχα. Τώρα, σαν τι οριακέ τιμέ, δεν έχει σημειωθεί ομοφωνία όσον αφορά το, το πού θα καθοριστούν αυτές οι οριακέ τιμές. Σε ποιο επίπεδο. Επίσης θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνει η κατάταξη σε διαφορετικές κατηγορίες ας πούμε μας είπε για, τα οχήματα σπορ ο εισηγητής. Καλά, εμείς θα να το εξετάσουμε. Τώρα για τα ηλεκτρικά και τα ευρυδικά. Θα πράθουμε τα πράγματα στο πλαίσιο τους. Θα πρέπει να δούμε τις διεθνείς προδιαγραφές για αυτά τα οχήματα. ένα πλαίσιο για να καλυφθούν αυτά τα οχήματα. Επίσης να υπάρχει κάποιος τόρυβος που να εκπέμπουν ελάχιστος αυτά τα οχήματα. Είναι καινούργια εφεύρεση, οπότε ακόμα δεν έχει διαμορφωθεί η κατάσταση όσον αφορά αυτόν τον θόρυβο. Το τελευταίο που θα είναι το εξή. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση όπως επανειλημμένα ανέφερε ο και οι Ναι, ξέρουμε ότι κάτι τέτοιο θα είναι σωστό και γι' αυτό ήδη έχουμε εγκρίνει κανονισμό για το θόρυβο των ελαστικών των αυτοκινήτων. έχουμε μεταβατικέ διατάξει με, θα ακολουθήσει η εφαρμογή, Επομένω ακόμα δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε εκείνον τον κανονισμό. Πάντως έχουν δρομολογηθεί εξελίξεις και άλλο τώρα, όσον αφορά τη διαβούλευση, υπενθυμίζουμε ότι αυτή η πρόταση δεν γεννήθηκε χτες. Εδώ και μια τριετία κυκλοφορεί, συζητείται, προετοιμάζεται στα διεθνή φόρα. Κάρτ 21 ανέφερε κάποιο, ε, αυτό, αυτό τον φορέα αυτοκινητοβιομηχανιών, με του οποίου ήρθαμε σε επαφή. Είχαμε διμερεί επαφέ. Και φυσικά κάναμε και την μελέτη των επιπτώσεων. Βάσει πάρα πολύ ενδελεχούς μελέτες για τα υπάρχει και τα κατά της ρύθμισης. Αυτό πρέπει. Σα ευχαριστώ πολύ που ήσασταν όσο γινόταν πιο σύντομο, Κύριε Παγνιό, θέλετε κάτι να πείτε. Ναι, Πρόεδρε, κοιτάω το ρολόι εργός και σα ευχαριστώ που είπατε ότι όντω τι τελευταίε εβδομάδε είχαμε το, πολύ σημαντικέ εκλογέ στη Γαλλία που όσο με αφορά είχε αίσιο πέρα, αλλά φυσικά αγαπητέ Ντομινίκ, τι να κάνουμε, εναλλαγή. Ε, και ήμουν όντω πολύ απασχολημένος. Πάντως σίγουρα θα συναντηθούμε με τους Σκιώδης τις επόμενες μέρες, ώστε να μπορέσουμε πριν τι 15 Μαΐου να υποβάλουμε αυτή την ενδεχομένω κοινή πρόταση και είδα ότι σε σχέση με τις διάφορες παρεμβάσει ότι υπάρχουν κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις κυρίως όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Κομισιόν αλλά θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να φτάσουμε σε συμβιβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πάρνιο. Να επαναλάβω την ε, προθεσμία για υποβολή τροπολογιών είναι 15η Μαΐου, η ψηφοφορία στην Επιτροπή Μεταφορών θα είναι τον Ιούνιο και η ψηφοφορία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, είναι για τον Ιούλιο. Και όπως ακούσαμε, ο εισηγητής θα συγκεντρώσει τους σκιώδης. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενο θέμα στη μερισσία διαταξή τώρα είναι το πακέτο ακρόασης για τα ε, αερολιμένες. Θυμάζομαι τον κύριο είναι εδώ. Είναι εδώ. Yeah, it's Matthew here? Matthew Walden.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 Okay, colleagues. Λοιπόν, συνάδελφοι. Περνάμε τώρα στο θέμα που αφορά το πακέτο των αεροδρομίων. Θα θυμάστε, σήμερα το πρωί ζήτησα πειθαρχία και ερωτήσεις, όχι ομιλίες το ίδιο επαναλαμβάνω και τώρα γιατί όπως βλέπετε το απόγευμα είναι ε, ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Υπάρχει και το ζήτημα των μελλοντικών ακροάσεων, θα τα δούμε. Αυτά με τους συντονιστές. Γιατί ε, υπήρξαν παράπονα ανθρώπους που δεν είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν και είναι δύσκολα τα πράγματα, πιστέψτε με. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε με τα γενικά του πακέτου αυτού με τον κύριο Baldwin. Ο κύριος Baldwin από τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Μετά θα πάμε στο πάνελ για τα slots, τα, τις χρονοθυρίδες και μετά θα περάσουμε στους περιορισμούς του θορύβου. Ακούσουμε τώρα τον κύριο Μπόλτγουν λοιπόν. Πέντε λεπτά έχετε. Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι γρήγορος και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσω το πακέτο των αεροδρομίων. Θα είμαι σύντομος, θα μείνω μέχρι το τέλος της ακρόασης και ε, ελπίζω να απαντήσω σε ερωτήσεις και τυχόν ανησυχίες. Δεν θέλω μόνο να σας πω το βασικά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα γιατί έχουμε αυτό το πακέτο. Πρώτα και, και κατά κύριο λόγο για λόγους πολιτικής. Τα ξέρετε. Τα αεροδρόμια έχουν σημασία, ε, προσφέρουν ανάπτυξη και δουλειές, είναι η πύλη της Ευρώπης στον υπόλοιπο κόσμο και εξυπηρετούν μεγάλο κομμάτι ε, της παγκόσμιας αεροπορικής αγοράς η Ευρώπη. Είναι το 1 τρίτο έχουν προκλήσεις. Πρώτον, δυναμικότητα. Αν δείτε τα πιο γρήγορα αναπτυσσόμενα αεροδρόμια, το 2010 ε, ένα από αυτά μόνο είναι στα ταχύτερα αναπτυσσόμενα του κόσμου. Το ότι έχουμε τρία στα δέκα κορυφαία γενικώ σημαίνει πως οι άλλοι σιγά σιγά καλύπτουν τη διαφορά. Αυτή τη στιγμή 19 αεροδρόμια μας θα έχουν φτάσει στα όρια τους το 2030 και έτσι περιορίζεται η συνεισφορά της ε, αεροπορίας στην ανάπτυξη της Ευρώπης και δεν θα είναι αποτελεσματικός ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός. Μετά έχουμε ζήτημα ποιότητας και ανταγωνιστικότητας. Ξέρω πως το ακούτε κάθε μέρα εδώ πέρα από τους χρήστες, δηλαδή τους επιβάτες. Έχει γίνει κάποια πρόοδος, αλλά ε, πρέπει να ε, γίνει περισσότερο. Αυτή είναι η λόγη της πολιτικής. Αλλά υπάρχει και ένα θέμα διαδικαστικό. Εμείς μετά από δική σας πρόταση κύριε Πρόεδρε ε, το κάναμε αυτό. Είχαμε τις προτάσεις του 2007 που έλεγαν πως δεν υπήρχε η απαραίτητη δυναμικότητα και τόνιζε τα βήματα που έπρεπε να ληφθούν. Η The Jensen Report για τις για η έκθεση Τζένσιν για την εξυπηρέτηση εδάφους ε, έλεγε πως έπρεπε να δούμε την ερμηνεία ορισμένων διατάξεων και γρήγορα να διευκρινίσουμε τις διατάξει που αφορούν την προστασία των εργαζομένων. Οπότε δεν ε, το κάναμε επειδή το θέλησαμε εμείς. Για τα slots. Όταν εμείς προτείναμε να σταματήσει ο κανονισμός ε, user προσωρινά, μας πιέσατε να κάνουμε μια αξιολόγηση αντικτύπου. Εμείς θεωρούμε πως θα μπορούσαμε να... και η έκθεση έλεγε πως θα μπορούσαμε να έχουμε κάποια στοιχεία αγοράς στον τομέα αυτό. Οπότε προσπαθούμε να αντιδράσουμε σε αυτά τα οποία ζητάει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ελπίζω οι προτάσεις μας να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας. Για τις προτάσεις τώρα αυτές σύντομα για τις φρονοθύλιδες στα αεροδρόμια δεν χρησιμοποιούνται όπως θα έπρεπε. Γι' αυτό προσπαθούμε να προωθήσουμε κινητικότητα των σλότς ε, μέσω μιας ε, εμπορευσιμότητάς τους σε μια δευτερογενή αγορά. Η δευτερογενής αγορά λοιπόν ε, θα διασφαλίσει πως θα πάνε τα σλότ σε εταιρείες που μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Η δευτερογενής αγορά επίσης σημαίνει πως θα υπάρχει και πιο ξεκαθαρή πληροφόρηση για το ποια σλότς είναι διαθέσιμα σε ποια αεροδρόμια. Και ένα άλλο σημείο βέβαια αφορά την ανεξαρτησία των συντονιστών που παίζουν μεγάλο ρόλο για την αποτελεσματική κατανομή τους. Και κάτι άλλο προκαλεί πολλές συζητήσεις εντός του Κοινοβουλίου. Προτείναμε να αλλάξουμε την αναλογία του κανόνα είτε το χρησιμοποιείς είτε το χάνεις σε ένα λόγο 85-15. Αλλά ε, ευχαρίστως να συζητήσουμε και να μιλήσω περισσότερο κύριε Πρόεδρε, αλλά θα ήθελα να παρακαλέσω το Κοινοβούλιο να αντισταθεί στο lobbying που υπάρχει. Είναι κατανοητό και φυσικό θα έλεγα κιόλας οι ενδιαφερόμενοι να προσπαθούν να προωθήσουν τις υφιστάμενες εταιρείε. Έχουμε όμως ταυτόχρονα καθήκον οι κανόνες να είναι αποτελεσματικοί και δίκαιοι για την εξυπηρέτηση εδάφους. Είναι σαφές, πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση και από πλευρά ποιότητα και αποτελεσματικότητα. Αλλά όπως και για τα σλότς αυτό το οποίο θέλουμε είναι εξέλιξη και όχι επανάσταση. Ε, στα λίγα αεροδρόμια που υπάρχει ακόμα επιλογή εταιρεία για τις αεροπορικές εταιρείε, μπορούμε να πάμε από δύο σε τρεις εταιρείε. Δεν θεωρούμε πως η προσεκτική αυτή αύξηση θα οδηγήσει σε πτώση της ποιότητας. Επίσης, δεν θεωρούμε πως αυτό μπορεί να είναι μια δογματική ε, πρόταση για περισσότερο ανταγωνισμό. Προτείνουμε και ποιοτικά κριτήρια κατόπιν πρόταση του Κοινοβουλίου. Και, πιο σημαντικό, βασικό σημείο της πρότασής μας είναι να διευκρινίσουμε το τι μπορούν να κάνουν τα κράτη-μέλη από τους κανόνες μας για να ενισχύσουν ε, τους κανόνες απασχόλησης όσων εργάζονται σε αυτόν τον κανόνα. Πρέπει να μπορούν να επιβάλλουν κανόνες στα κράτη-μέλη σε περιπτώσεις όπου η πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές είναι περιορισμένη. Επίσης υποστηρίζουμε την ελάχιστη ε, εκπαίδευση προσωπικού. Θεωρώ λοιπόν πως η πρότασή μας είναι δίκαιη και θεωρώ ισορροπημένη. Τέλος, λίγα λόγια για το θόρυβο. Και πάλι η λέξη ισορροπία εδώ πέρα ε, είναι πάρα πολύ σημαντική σε σχέση με το τι προτείνουμε για να ακολουθήσουμε την προσέγγιση του ΙΚΑΟ. Επίσης, είναι ισορροπημένη στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Όλοι θέλουμε να διασφαλίσουμε Λογικό είναι να προστατεύουμε τους πολίτες μας από τον υπερβολικό θόρυβο των αεροπλάνων. Ειδικά αυτούς που ζουν κοντά στα αεροπλάνα, αλλά νομίζω πως ε, πρέπει να λαμβάνονται προσεκτικά αποφάσει που έχουν τεράστιες επιπτώσεις. Εμείς λοιπόν δεν θα προτείνουμε παρά μόνο διαδικασίες οι οποίες πρέπει να γίνονται σεβαστές για τη λήψη αποφάσεων. Για να μην ε, λοιπόν παρεξηγηθώ. Σεβόμαστε πλήρως τη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Δεν έχουμε καμία επιθυμία, καμία όρεξη να λάβουμε τη μία ή την άλλη απόφαση επί της ουσίας. όσον αφορά του περιορισμού στο ρυθμό Αυτό το οποίο προτείνουμε είναι μέτρα για να αυξηθεί η διαφάνεια της διαδικασίας. Και υπάρχει ένα αποπτικό ρόλο για την Κομισιόν όσον αφορά τη διαδικασία, όχι την ουσία. Δεν επηρεάζονται εδώ πέρα οι στόχοι των κρατών μελών, δεν επηρεάζεται η ουσία των αποφάσεων και θεωρούμε πως η πρόταση σέβεται πλήρως την επικουρικότητα. Και πάλι σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου, εκπληρώνουμε και τις απαιτήσει της συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Οπότε θα μπορέσουμε να πιέσουμε τις ΗΠΑ για το άνοιγμα της αγοράς όσον αφορά την ιδιοκτησία. Έφτασα τα πέντε λεπτά και τα ξεπέρασα κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Για να ολοκληρώσω. Το πακέτο αυτό έχει στόχο καλύτερα αεροδρόμια και καλύτερη αεροπορία. Σε λιγότερο από τρεις μήνες λοιπόν στο Συμβούλιο υπάρχει ένας κοινό τόπος, μια βάση συνεννόησης για δύο βασικά ζητήματα, πρόσβαση και προστασία των εργαζομένων. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για τον θόρυβο και τα σλότς. Καλώς ορίζουμε τη σημερινή ακρόαση ω ένα πολύ σημαντικό μήνυμα της πρόθεσης του Κοινοβουλίου να προωθεί αυτό το ζήτημα. Σα ευχαριστώ για τον χρόνο και την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κύριε Μπόλτουιν. Ο κύριος Μπόλτουιν θα φύγει τώρα από εδώ, αλλά μην ανησυχείτε. Ε, δεν θα φύγει από την αίθουσα. Απλά δεν ε, φτάνει το έδρανο εδώ του Προεδρείου για όλους ε, τους προσκεκλημένους τα καθίσει εκεί πέρα, στα έδρανα της Κομισιόν. Οπότε, σκοπεύω οι Ούγες Σασάουι και Λάιχτφριντ, οι εισηγητές, να ακούσουν τους εμπειρογνώμονες και μετά να ακούσουμε εσάς τους εισηγητές στο τέλος ε, για να μας πείτε τα δικά σας και ίσως να συνοψίσετε τα πράγματα. Αν συμφωνείτε. Ο κ. Λάιχτφριντ δεν έχει έρθει. Νομίζω οι υπόλοιποι δύο συμφωνούν. Οπότε, μπορούμε να περάσουμε στον πρώτο ομιλητή για, ε, για πέντε λεπτά. Έχουμε τον Σάιμον Σμιθ από την Steer Ντέιβις Κλίβ, συντάκτης της αξιολόγησης αντικτύπου. Να σας πω πως ποτέ πριν στην ιστορία του Κοινοβουλίου δεν είχε προκαλέσει μια συζήτηση τόσες ε, συζητήσεις. Έχετε λοιπόν τον λόγο κύριε Σμιθ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάντα σας δώσω το ιστορικό πλαίσιο, διότι ήδη αναφέρθηκε ότι ε, πάρα πολλά ε, έχουν πια γεμίσει, έχουν καργάρει 3-4% είναι η αύξηση της κυκλοφορίας και, και βέβαια δεν γίνεται να, να επεκτείνουμε τα αεροδρόμια. Ε, θόρυβος, μόλυνση. Οπότε όλο ένα και περισσότερα από αυτά βρίσκονται σε σημείο κορεσμού και να, όπως είναι για το χήθρο. Άρα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις ε, χρονοθυρίδες. Δεν, λέμε θα λυθεί το πρόβλημα της, της ε, αλλά θα, πρέπει να τις εκμεταλλεύουν για ρυθμίσεις όσο γίνεται καλύτερα. Εδώ πέρα έχουμε διάφορες γραφικές παραστάσεις όσον αφορά την, ε, τη, τη ζήτηση και το πώς γίνεται η κατανομή, αφορά το αεροδρόμιο της Βιέννης και το Χήθρο είπαμε ότι όλο ένα και περισσότερα αεροδρόμια έχουμε σαν το Χίδρο, οπότε ε, έχουμε τέτοιου είδους κατανομή και οι χρονοθυρίδες ε, πιάνουν όλη, όλη την, την, την ημέρα στις εργάσιμες ώρες, οπότε δεν υπάρχουν κενά στο σύστημα. Το ισχύον τώρα σύστημα ε, είναι διοικητικού, διεκπαιρεωτικού χαρακτήρα. Οι αεροπορικές εταιρείε έχουν ιστορικά δικαιώματα ε, αρκεί να πληρούν κάποια περιορισμένα κριτήρια, δηλαδή χρησιμοποιήσει το σλότ ή το χάνει είναι ο βασικός κανόνας. Είναι δύσκολο ένα ανταγωνιστής να τρυπώσει ε, σε τέτοια, σε τέτοια κατάσταση ε, ανταγωνισμού. Η Ryanair, η Jeter τελικά μπόρεσαν να αναπτυχθούν εκτός αυτών των κορισμένων αεροδρομίων σαν τη Φραγκφούρτης ή του χύθρου οι αεροπορικέ εταιρείε επομένως έχουν αυτά τα σλότ για ιστορικού λόγους, διότι 10-20 χρόνια βρίσκονται στην αγορά, αλλά τελικά όμω δεν είναι αναγκαστικά αυτέ οι ιστορικές εταιρείε οι πιο αποτελεσματικέ στη χρήση. Το θέμα είναι ότι εάν έχουμε κάποιο μηχανισμό τη αγορά ε, θα έπρεπε να γίνεται κάποιο είδου εμπόριο και αυτό σημαίνει ότι αυτοί που έχουν τα πιο μεγάλα αεροπλάνα, πιο πολλούς επιβάτες, αυτοί που λειτουργούν ε, ε, όλο το χρόνο και όχι μόνο στις περιδεχνείς, ε, τότε θα είχαμε και κριτήρια αεροδρομίου όπως η Φραγκφούρτη, το Χίθρο και οπότε θα πρέπει να δούμε το πώς θα γίνει πώς θα γίνεται αυτό το η συναλλαγή, αυτό το εμπόριο των χρονοθερίδων. Πάντως δεν μπορεί να γίνει με κάποιο πληστηριασμό. Δεν είναι πρακτικό στις περισσότερες περιπτώσεις. Επίσης έχουμε κάποιο δευτερογενή αγορά των σλότς ε, το οποίο ούτε το απαγορεύει ούτε το προβλέπει ρητά η ισχύουσα νομοθεσία. Και εάν και ε, επεκταθεί αυτού του είδους δευτερογενή αγορά θα μπορούσε να βοηθήσει τα κόρεσμενα αεροδρόμια και μακροπρόθεσμα θα βοηθήσει γιατί όλο ένα και πιο πολλά αεροδρόμια γίνονται περισσότερο κορεσμένα. Και η ανάλυση μας λέει ότι με δευτερογενή αγορά θα έχουμε όλα τα υπέρ τους προτινομένες δέσμες μέτρων. Άλλες προτάσεις τώρα είναι οι εξής. Όπως προείπαμε, η κατακύρωση, ας το πούμε, η κατανομή θα πρέπει να γίνει τόσο πιο αποτελεσματική και τα μέτρα που θέλουν να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική χρήση από τις αεροπορικές εταιρείες διαφάνεια στα δεδομένα, προς κάθε κατεύθυνση κλπ. Και κάποιες μικρές αλλαγές μπορούμε να επιφέρουμε, ούτως ώστε να ε, μπορέσουμε να έχουμε ε, ρύθμιση και κάλυψη περισσότερων, ε, περισσότερων πτήσεων, όπως ας πούμε το, το, το, αν έχει, να αξιοποιούνται πλήρω και σε όλη την ημέρα η, τα σλότς ακόμα και αυτά που έχει κανεί καθυστερήσει να αξιοποιήσει. Όμως, χρειάζεται να αποφασίσει κανείς ποιες εταιρείες θα καλυφθούν και ποιες δεν θα καλυφθούν από αυτές τις ρυθμίσεις. Βεβαίως, Δεν μπορούμε να καλύψουμε τα πάντα και θα πρέπει να γίνει κάποιο είδους ε, αντιστάθμιση σε σχέση με το κάποιες εφορικές υπηρεσίες πρέπει να καλυφθούν και κάποιες να μείνουν απ' έξω. Ευχαριστούμε Σάιμον, ο Πρόεδρος. Πάμε Μόργαν Φούξ, από την ACI Morgan Φούξ, διευθυντής στην ε, ACI, στον φορέα για τα διεθνή αεροδρόμια. Ευχαριστούμε που μας, μας καλέσατε. Που να σας πω ε, ότι έχουμε, ότι εκπροσωπούμε 350 αεροδρόμια 6 χωρών. Όταν συζητήσαμε αυτό το κείμενο, προσπαθήσαμε να λάβουμε υπόψη τι θα γίνει στα αεροδρόμια στο μέλλον. Πάρα πολύ καλά τα διατύπωσε η Επιτροπή. Έλαβε υπόψη πολλά στοιχεία της δέσμης μέτρων. Καλή ανάλυση όσον αφορά το πώς θα επηρεάσει τις αεροπορικές μεταφορές στην Ευρώπη αυτό το, το, αυτό το μέτρο. Το 2030 θα έχουμε διπλασιασμό της κυκλοφορίας και θα, έχουμε πολύ περισσότερο τρόπο που θα, θα έχουν κορεστεί σαν το χύθρο. Επομένως δεν τα πάμε πάρα πολύ καλά όσον αφορά το να μπορέσουμε να καταφέρουμε τις δυνατότητές μας γιατί χρειάστηκαν 15 χρόνια τόσο ώστε να, μπορέσουμε να, πούμε, να κάνουμε ένα καινούριο διάδρομο προς γύρω στη Φραγκφούρτη και να μπορέσουμε να καλύψουμε και τις νυχτερές πτήσεις και στο Μόναχο, στο Χίθρο τώρα που θα δούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, άρα θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε καλύτερα τι δυνατότητε των αεροδρομίων και εγκαίρω τόσο ώστε να καλύψουμε κάθε φορά τη μέλου ζήτηση. Οπότε αυτό θα βεβαίω είναι ε, αρμόδια των κρατών μελών, αλλά θα πρέπει να αξιοποιήσουμε πλήρω την υπάρχουσε δυνατότητε δυνατότητα και περί αυτού πρόκειται εδώ στην πρόταση τη Επιτροπή. Δεν λέμε να αρχίσουμε από το Α, να τα γκρεμίσουμε όλα και να τα χτίσουμε την αρχή. Απλώ θα πρέπει να δούμε τι γίνεται, να μην έχουμε ε, κατάσχεση επίσχεση των πρώτων των σλότς και εδώ πέρα τα λέει καλά η Κομισιόν, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία σε του τους κανόνες προσαρμογής στις τοπικές ε, ανάγκες αγοράς και να δούμε ποιος είναι ο ρόλο του διαχειριστή δικτύου, Network Manager. Επίσης ε, θεωρούμε ότι μια σειρά προτάσεων της Επιτροπής σίγουρα θα βελτιώσουν την αξιοποίηση των σημερινών δυνατοτήτων όπως την νομιμοποίηση της δευτερογενούς αγοράς ε, ε, να τροποποιηθεί ο κανόνας του νεοεισερχομένου να γίνει λιγότερο υποχρεωτική ρύθμιση και έτσι να βοηθεί ο ανταγωνισμός, περισσότερη διαφάνεια γενικά όσον αφορά την επιδίκαση, κατακύρωση των σλότς από 80 στα 20 να πάει στο 85-15 ο λόγος, η αναλογία χρήσης Και έτσι να έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία, να καλύψουμε ανώτερα βία, ε, απεργίες κλπ. Γιατί είναι θεμητό που να θέλουν και οι οδηγίες και οι εταιρείε, συγγνώμη, να χρησιμοποιήσουν δυνατότητες που δίνονται όσο γίνεται περισσότερο. 15 τα σλότς που θέλει ο καθένας μέσα στη μέρα, σε καλοκαίρια, χειμώνα, ε, κατά πόσο θα είναι ε, στη σειρά, ε, η μία μετά την άλλη, μετά την άλλη, διακοπτόμενα τα σλότς που δίνονται και επίσης να εξασφαλιστεί γενικότερα ευελιξία και για τα αεροδρόμια και για τις ευρωπαϊκές εταιρείε ούτω ώστε οι σημερινές δυνατότητες να αξιοποιούνται τώρα. Πιο συγκεκριμένα, να ρίξω μια ματιά σε κάποιες από τις επιπτώσεις της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, έχουμε εδώ μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα. Για παράδειγμα έχουμε αύξηση του κανόνα 80-20 σε, σε 85-15 όπως για τον και όταν υπάρχει ένας μονοδιάδρομος. Όμως πήγαμε σε, σε εκατομμύρια, 60 εκατομμύρια και πάμε στο 85% ε, και έτσι θα έχουμε 320 επιπλέον πτήσεις ή σλότς που θα χρειαστούν το καλοκαίρι. Γι' αυτά μέχρι το 2007, δηλαδή 320 παραπάνω σλότ θα μπορούσαν να πάνε πίσω και να ξαναγυρίσουν προς ανακατανομή. Αντίστοιχα, θα δούμε τι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν αυξηθούν από 5 σε 15 εβδομάδες οι σειρές των σλότς, αυτό σημαίνει ότι θα πάμε σε 371 πλέον ε, ε, πτήσεις που θα μπορούσαν να έχουν γίνει στον Κάτουικ. Τώρα, για την κράτηση, για τις ε, κρατήσεις, το μπλοκάρισμα. Στον Τίρφεντ ε, αυτό, ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2002 και για τέσσερα χρόνια και αποτέλεσμα ήταν η μείωση των μη εκμεταλλευθέντων σλότς. σλότς Και εγκατακλείδη, στον 10% μειώθηκε και άρα έτσι θα έχουμε πιο αποτελεσματική χρήση. Άρα θα πρέπει να δούμε τι νομοθετικές προτάσεις θα γίνουν, γιατί νομίζουμε ότι έτσι θα έχουμε καλύτερη εξορρόπηση των συμφερόντων, από τη μία των αεροδρομίων και από την άλλη των ε, εταιριών. Σας ευχαριστώ. Νομίζω πως θα αλλάξετε θέση τώρα με τον κύριο Καν για να έχει και αυτός πρόσβαση στο μόνο λάπτο που υπάρχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. So the next Επόμενος ο ο κύριος Ατάρ Χουσέιν Χάν από την Ένωση ε, Ευρωπαϊκών Αεροπορικών Εταιριών. Έχετε το λόγο για πέντε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ πέρα σήμερα και μπορώ να αναφέρω τις απόψεις της ε, Ένωσής μας. Να σας υπενθυμίσω πως εκπροσωπούμε 34 αεροπορικές εταιρείες, γύρω στις 11.000 πτήσεις τη μέρα και μιλάμε και για διυπηρωτικές πτήσεις και ευρωπαϊκές, οπότε αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα αυτό σε ολόκληρον κόσμο σε καθημερινή βάση ενδιαφέρον είναι πως ο τίτλος είναι πως να αυξηθεί η δυναμικότητα των αεροδρομίων. Να σας πω πως ο κανονισμός των σλότς είτε με την τωρινή του μορφή ε, δεν θα αυξήσει την ε, δυναμικότητα των αεροδρομίων. Η δυναμικότητα των αεροδρομίων αυξάνεται με το να φτιάχνουμε αεροδρόμια, υποδομές. Βλέπουμε εδώ πέρα δύο πόλεις Ευρώπης, Λονδίνο και Φραγκφούρτη, που φιλοξενούν μεγάλα αεροδρόμια της Ευρώπης σε σχέση με το τι συμβαίνει στην Κίνα και τη Μέση Ανατολή. Και θα εκπλαγείτε από το γεγονός πως στο Ντουμπάι, όπου ο αριθμός των επιβατών μεταξύ τώρα και το 2020 θα αυξηθεί από, 16, από 60 εκατομμύρια σήμερα σε 260 εκατομμύρια σε 10 χρόνια. Αυτή την παρατηρήση έχω να κάνω. Το να αυξάνουμε την δυναμικότητα των αεροδρομίων είναι απλό περισσότερες υποδομές. Δεν έχει σχέση με τα σλότ. Θα περάσω αυτή τη διαφάνεια. Πάμε σε αυτήν εδώ. Το σύστημα κατανομής σλότ. Είναι παγκόσμιο, όπως ξέρετε. Όταν πηγαίνει κάποιος από το αεροδρόμιο Α στο αεροδρόμιο Β ε, και, και τα δύο περιορίζονται από σλότ. χρειάζεται κανείς δύο ε, σλότ. Ε, αναχώρησης και άφηξης. Οι κανόνες λοιπόν πρόσβασης πρέπει να είναι οι ίδιοι και στις δύο άκρες και στο αεροδρόμιο αναχώρησης και αύξησης δεν έχει νόημα να είναι διαφορετικοί οι κανόνες. Και το ερώτημα είναι το εάν η Ευρώπη πάλι θα προσπαθήσει να κάνει δικούς της κανόνες. Επειδή εγώ είμαι από τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείε, πρέπει πω δεν είναι πολύ καλή ιδέα αυτό. Μεγαλύτερη διαφάνεια. Έχουμε πει πολλές φορές πως θεωρούμε πως χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια στον κανονισμό και μας ενθαρρύνει το ότι η Κομισιόν το είδε αυτό και σε σχέση με την διαφάνεια των συντονιστών και σε σχέση με τη διαφάνεια της διαδικασίας ε, για το δευτερογενές εμπόριο και πάντα λέγαμε πως ε, όσοι βεβαίω είναι κακοήθης θα πρέπει να τιμωρηθούν και υποστηρίζουμε οποιοδήποτε τέτοιο μέτρο. Η αρχή τώρα του κανόνα 80-20, είτε το χρησιμοποιείς ή το χάνεις. Βλέπουμε πως αν υπάρχουν σλότ σε 10 εβδομάδες έχουν την δυνατότητα οι αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν δύο από αυτές. Το να πάνε στο 85-15 κατ' ουσίαν σημαίνει πως θα είναι σε θέση να ακυρώσουν μία από τις 10 πτήσεις. 85-15 τι σημαίνει κατ' ουσίαν. 90-10. Έτσι. Και είναι αδύνατο για τις εταιρείε για οποιονδήποτε παράγοντα κάτι συνέβη, η συντήρηση αεροσκάφους, ε, ανωτέρα βία, να ακυρώσουν μια πτήση. Και δεν μπορούν έτσι να κρατήσουν τα σλότ τα οποία έχουν. Κάτι το οποίο τους δίνει κίνητρο να λειτουργούν μόνο και μόνο για να διατηρήσουν το σλότ. Κάτι το οποίο δεν στέκει ούτε οικονομικά και δεν νομίζω πως χρειάζεται να σας πω τι κάνει στο περιβάλλον. Αντιλαμβάνομαι πως από τη σκοπιά του αεροδρομίου μπορεί να πούν πως είναι αποτελεσματικό το αεροδρόμιο να αυξήσει τη χρήση του σε ολόκληρη τη σεζόν. Αλλά εάν είναι αποτελεσματικό το... Είναι αποτελεσματικό όμως και για την αεροπορική εταιρεία. Τώρα, να αυξηθεί η σειρά των σλότ. Ο Μόργαν είπε γιατί είναι υπέρ τα αεροδρόμια. Εμείς διαφωνούμε. να αυξηθεί ο κανονισμός, ο ορισμός με της σειράς των σλότ δεν αυξάνει τη δυναμικότητα. Στην πάνω γραμμή βλέπετε το τωρινό σύστημα όπου έχουμε τρεις αεροπορικές εταιρείες πολύ στριμωγμένες και έτσι ε, έχουμε τη μεγιστοποίηση της δυναμικότητας. Στο δεύτερη σειρά βλέπετε τον ορισμό των 10 διαδοχικών υποχρεωτικών εβδομάδων και θα υπάρχει μία εβδομάδα από τις 21 η οποία δεν θα χρησιμοποιείται και γίνονται ακόμη χειρότερα τα πράγματα αν δείτε την τρίτη γραμμή όπου αν επιλέξει μία εταιρεία να λειτουργήσει κάπου στη μέση αυτών των 21 εβδομάδων δηλαδή ουσιαστικά πριν και μετά από αυτές δεν υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας για άλλες εταιρείες. Και το ίδιο βλέπετε μπορούμε να πούμε και για την θερινή σεζόν που είναι 31 εβδομάδες τα πραγματίδια, απλά μιλάμε για α, περισσότερες εβδομάδες. Τώρα, τα τέλη κράτησης του σλότ. Πέρα από αυτά τα οποία πληρώνουν τα τέλη αεροδρομίου οι εταιρείε, συχνά προχρηματοδοτούν την ε, υποδομή πριν τη χρησιμοποιήσουν. Το ζήτημα είναι εάν χρειάζεται και τέλος κράτησης ή ακύρωσης. Ήδη υπάρχουν πολλές διατάξεις για τις κυρώσεις όσον αφορά την περίπτωση ακύρωσης της πτήσης. Το ερώτημα είναι ποιο θα είναι το κόστος, ποιος θα το πληρώσει και τέλος αντιβαίνει τον κανόνα 80-20 που όπως είπα επιτρέπει 20% ακυρώσεων και ακόμα και αν αυξηθεί στο 85-15 δηλαδή κατ' ουσίαν 90-10 πάλι ισχύει αυτό που σας είπα. Τελευταία διαφάνεια αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε και θα τελειώσω. Τα αεροδρόμια, τα δικτυωμένα που υπάρχουν εδώ πέρα στην πρόταση είναι μια έννοια λανθασμένη. Ο νέος ευρωπαϊκός ουρανός έχει διαχειριστεί δικτύου και αυτός λέγεται Eurocontrol που ε, ασχολείται με την πρόβλεψη και διαχείριση των ροών του δικτύου. Εμείς δεν θεωρούμε πως χρειάζεται δεύτερο επίπεδο διαχείρισης δικτύου και θεωρούμε πως ο κανονισμός των σλότ δεν σχεδιάστηκε ποτέ για τη διαχείριση των δικτύων. Είναι ένα εργαλείο προγραμματισμού για μήνες μπροστά, όχι καθημερινής διαχείρισης. Τέλος, κοστίζει το να επεκταθεί αυτή η διαδικασία σε κάθε αεροδρόμιο στην Ευρώπη είναι υπερβολή που κοστίζει πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Καν. Ο επόμενος είναι ο κύριος Ρίτσαρντ Μάθιος που είναι επικεφαλής ε, των σλότς και του προγραμματισμού της EasyJet. Okay, okay, Mr. Matthews, is yours for five minutes. Έχετε το λόγο για πέντε λεπτά, κύριε Μάθιους. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλύτερα με μικρόφωνο. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι εδώ σήμερα εκπροσωπώντας την EasyJet. Είμαστε ευτυχείς που μας δόθηκε ευκαιρία ως αεροπορική εταιρεία να έρθουμε εδώ και να σας ε, μιλήσουμε, είναι μάλλον ε, καλό ε, το ότι εμείς ως αεροπορική εταιρεία είμαστε μια εταιρεία που έχει ωφεληθεί πάρα πολύ από το γεγονός ότι υπάρχει ο κανονισμός περί σλότ. Είμαστε από αυτές τις εταιρείες που θεωρούμε πως ο κανονισμός των σλότ έχει σχεδιαστεί για να δημιουργηθεί ακολουθούν και άλλες εταιρείες, γιατί είμαστε και σχετικά νέα αεροπορική εταιρεία, ωστόσο είμαστε η τέταρτη μεγαλύτερη, μεταφέρουμε πάνω από 55 εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως και αν και έχουμε έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν, είμαστε, δεν έχουμε ως επίκεντρο το Ηνωμένο Βασίλειο και βλέπουμε τον κανονισμό αυτό όχι από την πλευρά του Heathrow ή του Gatwick γιατί το 60% των επιβατών μας προέρχονται από αεροδρόμια εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου. Γι' αυτό και μας ενδιαφέρουν πολύ αεροδρόμια όπως αυτά του Παρισιού, τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Ισπανίας και πέρα από, αυτά, από αυτές τις χώρες. Γιατί πετάμε σε κάθε αεροδρόμιο, η Φραγκφούρτη και το Heathrow είναι τα μόνα αεροδρόμια στα οποία δεν πετάμε αυτή τη στιγμή, αλλά πιστεύω ότι όσον αφορά τα υπόλοιπα είμαστε σε κατάλληλη θέση ώστε να μπορούμε να αξιολογήσουμε τη δυνατότητά μας να μπούμε σε αυτές τις πολύ κορεσμένες αγορές. Έχουμε την κυρία Κάρολιν Μακόλ στην συμβουλευτική ομάδα του Επιτρόπου Μεταφορών. Τα, οι πτήσεις μας δεν ξεκινούν όλες από κεντρικά αεροδρόμια, αλλά οι περισσότερες ναι. Ε, και γι' αυτό είναι σημαντικό για μας να εξετάσουμε σοβαρά αυτό το κανονισμό και να εξασφαλίσουμε τη την θετική λειτουργία του για μας γιατί πετάμε και σε κάποια αεροδρόμια τα οποία δεν είναι κορεσμένα αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις πετάμε προς κορεσμένα αεροδρόμια και θέλουμε έναν κανονισμό που να λειτουργήσει καλά ε, για μας θετικά. Υπάρχουν πολλά στοιχεία του προτινόμενου κανονισμού που τα υποστηρίζουμε αυτό θα πρέπει να είναι σαφές. Σημείωσα κιόλας ότι έχουμε κάποιες ε, ε, αντιφάσκουσες απόψεις. Βέβαια, εξαρτάται από πού βλέπει κανείς, από ποια οπτική γωνία βλέπει κανείς ε, το θέμα. Θα μπορούσαμε να... Εμείς είμαστε υπέρ της, ε, του δευτερεύοντος εμπορίου των σλότ. Υπάρχουν κάποια αεροδρόμια που είναι πολύ κορεσμένα και ακριβώς λόγω ενό περιβαλλοντικού συστήματο ποσοστό που σημαίνει ότι δεν μπορούν να δημιουργηθούν περαιτέρω σλότζ, αν υπήρχε δευτερεύον εμπόριο, αεροδρόμιο όπω το, αυτά του Παρισιού, του Παρισιού, θα μπορούσαμε εκεί να έχουμε καλύτερη πρόσβαση ως EasyJet. Είμαστε υπέρ τη αύξηση του κατοφλίου για τι νέε εταιρείε. Σε πολλέ περιπτώσει, παλιότερα όταν ξεκινήσαμε δεν είχαμε πρόσβαση στα αεροδρόμια αυτά και κάποιες περιπτώσεις Όμω είμαστε πια η μεγαλύτερη εταιρεία όπω το Gatwick. Σε άλλα αεροδρόμια προσπαθούμε ακόμα να πιαστούμε γιατί υπάρχει πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Σε πολλά αεροδρόμια, αν ε, και έχουμε φτάσει στη δεύτερη θέση, εξακολουθούμε να έχουμε 5 ή 7% των σλότ, που δεν είναι μεγάλος όγκο για να μπορέσει να υπάρξει ε, ε, ε, θεμητός ανταγωνισμός για, όλες τις, για όλους τους προορισμούς με, τον βασικό, με τη βασική αεροπορική εταιρεία. Θέλουμε να φτάσουμε το 10%. Θα πρέπει ωστόσο να το υπολογίσουμε με βάση το ποσοστό, τον όγκο των σλότς που είναι διαθέσιμα και τον χρόνο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με βάση το συγκεκριμένο σύστημα του κάθε αεροδρομίου. Το 10% λοιπόν είναι πολύ καλό ήδη. Υπάρχουν κάποιοι τομείς, μάλλον άλλο σημείο είναι ότι εμείς είμαστε υπέρ της διαφάνειας των σλότ συνεργαζόμαστε με τους συντονιστές των σλότ στην Ευρώπη και δεν γίνεται πάντα κοινή εφαρμογή του κανονισμού γιατί κάποιο κομμάτι της ε, διατύπωσης αφήνεται σε ελεύθερη ερμηνεία και οι ερμηνείες διαφέρουν. Θα θέλαμε οι συντονιστές των σλότ να χρησιμοποιούν το ίδιο σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο να είναι πολύ προηγμένο, ώστε ο συντονιστής των σλότ να έχει τη δυνατότητα να βελτιστοποιήσει τη χρήση των σλότ. Θα θέλαμε λοιπόν να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια με στόχο να, στηριχθεί, να στηριχθούν οι συντονιστές των σλότ για να χρησιμοποιούν τα καλύτερα δυνατά συστήματα. Όσον αφορά λοιπόν τις ανησυχίες μας, να σας πω ότι βασικά έχουν να κάνουν με τις ε, μίνιμουμ ε, σειρές, δηλαδή την μείωση του λόγου από 80-20 σε 85-15 μπορούμε να έχουμε το κατόφλι 85% μόνο αν έχουμε μίνιμουμ ε, σειρά σλότ 20 εβδομάδων. Το 85% όμως δεν θα λειτουργούσε για το καλοκαίρι, ακόμα και για 15 εβδομάδες. Χρειάζεται μια σειρά 20 εβδομάδων για να μπορεί να έχει νόημα ένα τέτοιο ποσοστό. Γι' αυτό είπαμε ότι δεν υποστηρίζουμε την αύξηση από το 80 στο 85, γιατί στην ουσία, στην πράξη, δεν αντιστοιχεί σε κάτι συγκεκριμένο. Και ποιο άλλο πρόβλημα είναι αυτή η σειρά ε, των, του μάλλον το μήκο τη σειρά των σλότ. Τα σλότα ε, χορηγούνται με τη βάση εβδομάδων. 30 εβδομάδε το καλοκαίρι, 22 το χειμώνα, φτάνουμε στις 52 του χρόνου και αυτές τα, τα σλότ, τις σειρές των σλότ ε, χορηγούνται ε, με βάση αυτές τις ε, χρονικές περιόδους. Αν το γεγονός ότι ο Αύγουστος, ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος δήθεν ανήκουν σε διαφορετική εποχή είναι ένα ανόητο επιχείρημα. Στην ουσία η σεζόν είναι από τα τέλη Μαρτίου μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου το καλοκαίρι. Το θέμα κλειδί είναι ότι έχουμε πολλές, ε, πολλές προορισμούς όπου θα θέλαμε να λειτουργούμε 10 μήνες το χρόνο, Σεπτέμβριος μέχρι και τέλος Ιουνίου, αλλά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θέλουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Όπως συμβαίνει εδώ στις Βρυξέλλες, πολλές ε, εταιρείε κλείνουν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και είναι τρελό οι εταιρείε να συνεχίζουν να λειτουργούν με βάση ένα κανονισμό που τους αναγκάζει να πετούν τις ίδιες πτήσεις όπως τον Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο και μετά ξανά τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Μία σειρά λοιπόν 15 εβδομάδων δεν θα επέτρεπε σε, στις εταιρείε να πετούν Σεπτέμβριο-Οκτώβριο με διαφορετικό τρόπο από ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. όπου θα θέλαμε δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε τα αεροπλάνα μας για να κάνουμε πτήσεις αναψυχής και όχι business. Οι 15 εβδομάδες λοιπόν δεν αντιμετωπίζει το γεγονός ότι μπορεί κανείς να διακινδυνεύσει να χάσει τις, τα του, γιατί ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος είναι μόλις οκτώ εβδομάδες σειρά. Αυτά ευχαριστώ. Thank you very much Εμείς ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Ξαναλάζουμε θέσεις. Σαν το παιχνιδι αυτο αυτό, πάνε γύρω-γύρω για αλλάζουν κάθισμα. Ποιος θα μείνει Τώρα το επόμενο. Ωραία που εκπροσωπεί 36 Ιταλικά ε, αεροδρόμια ή 39 τέλος πάντων διαμετής στην Ιταλία πάντα είναι αυτά τα αεροδρόμια και αυτό το οποίο έχουμε απομένει είναι απλό. Θα πρέπει οι δέσμοι των ρυθμίσεων να καλύψει την ανάγκη εξυγχρονισμού, να υπάρχει συντονισμός αυτών των μέτρων. Το θέμα είναι τι προσδοκούν τα δικά μας αεροδρόμια. Ο στόχος, ο βασικός είναι να μπορέσουμε να προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες στην επιβάτη και έτσι ε, δίνεται η δυνατότητα του να εξελιχθούμε, να έχουμε πρότυπα ποιοτικά, πιο ισόρροπη προσέγγιση. Για να δούμε τώρα συγκεκριμένα το θέμα των χρονοθερίδων. Υπήρξε εκείνη δεύτερη δεύτερη για τον ε, Ευρωπαϊκό Ουρανό και θα θυμάστε ότι το θέμα ήταν το πώς θα διαχειριστούμε την ενέργεια κυκλοφορία. Ίσως ορισμένοι εξημών δεν γνωρίζετε ότι ε, εκείνη δεσμή έχει και έναν πυλώνα που αφορά τις υπηρεσίες εδάφους, τέλο πάντων τη διαχείριση των θεμάτων που γίνουν στο έδαφος και σε τουλάχιστον δύο νομοθετήματα μπορεί να δείτε τέτοια θέματα, ε, τέτοιες, τέτοιες επιχειρήματα για τις υπηρεσίες εδάφους και για το διαχειριστή δικτύου που ε, λέει για το πώς ο, tour operator, αυτή η, υπηρεσία, η επιχείρηση τουριστικών υπηρεσιών έχει να παίξει σημαντικό ρόλο, συντονιστικό και για να δούμε εμείς τι ρόλο μπορούμε να παίξουμε σε αυτό το σημαντικό πρόβλημα. Είναι η τουριστική επιχείρηση ε, κάποιος που έχει συντονιστικό ρόλο και αυτό έχει ρίζες στο παρελθόν. Μέχρι σήμερα το σύστημα λειτουργεί καλά. Να μην υποτιμούμε επίσης τον, τον ρόλο των αεροπορικών εταιριών στην, στο να λειτουργούν όλα αυτά τα συστήματα και τα, και, η και τα αεροδρόμια και οι χρονοθυρίδες και οι υπηρεσίες εδάφους. Επομένως θα πρέπει να δούμε ποιο ποια είναι η, η πιο ισόρροπη ρύθμιση που θα πρέπει να κάνουμε μεταξύ της ρύθμισης από πάνω ή από τη βάση να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες οι τοπικές. Και θα λαμβάνονται υπόψη και από τα κρατημέλη και από την Επιτροπή Συντονισμού. Συγγνώμη τώρα για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε κάποιες αλλαγές και κάποιες βελτιώσεις που μπορούμε να επιφέρουμε. Ας πούμε, το ποιες είναι οι παράμετροι που θα ρυθμίσουν την αντιμετώπιση. Να μην υπάρχει σύγχυση στο πώς θα είναι καλύτερη εξισορρόπηση. Οι εμπλεκόμενοι μας συμμετάσχουν πλήρως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι ε, επίση και οι διαχειριστές ε, δικτύου, ενδεχομένω να συμμετέχουν ως παρατηρητές. Πρόκειται για λειτουργικό χαρακτήρα μέτρο. Και επίσης να μην έχουμε δυσμενείς διακρίσεις, αλλά να έχουμε διαφάνεια. Το αξίζουν αυτό οι τουριστικές επιχειρήσεις και οι αεροπορικές εταιρείε. Ξέρουμε τι κυρώσεις έχουν επιβληθεί για την άσκηση των οικονομικών αυτών δραστηριοτήτων το βράδυ θα πρέπει να δούμε το ότι ίσως δεν είναι οι Βρυξέλλες ε, η μοναδική πηγή ρύθμισης του κλάδου. Επίση, ε, για το πώς μπορεί να ρυθμιστούν τα προβλήματα, λάβετε υπόψη σαν παράδειγμα το αεροδρόμιο Λινάτε του Μιλάνου. Είναι κορεσμένο και κάποια στιγμή λήφθη κάποια απόφαση από τα πάνω. Όμως, δεν είναι μόνο το Λινάτε. Έχουμε και το Μαλπένσα και το αεροδρόμιο του Μπέργαμο. Ιδίω το Μαλπένσα είχε, το, το είχε το κοινοβούλιο και άλλα θεσμικά όργανα υπό την αιγίδα τους. Και έχουμε και πολλές δυνατότητες που μπορούμε να αξιοποιήσουμε στο Μαλπέντσα. Πολύ ενδιαφέρουσα η απόφαση των αρχών αντιτράστ, ούτως ώστε να έχουμε μια υποκατάσταση του νοσοδρομίου με το άλλο. Και έτσι ε, αυτό αφορούσε τις συνδέσεις, όλες τις συνδέσεις εκτός από Μαλπέν, Σαλινάτε, Ρώμιο. Αν έχουμε συνδυασμένους τρόπους μεταφοράς, τότε κανείς κάνει τη διαφορά όσον αφορά την αξιοποίηση των δυνατήτων. Όπως και άλλες χώρες, και στην Ιταλία υπάρχει πρόβλημα δημοσιονομικό. Όμως τα τέλη αεροδρομίων έχουν παγώσει στην Ιταλία για πάνω από 10 χρόνια. Έγινε, μόνο, γίνεται μια μικρή άτα επιβάλλεται. Κατά μέσο όρο παίρνει 10 χρόνια για να κάνουμε μια επένδυση πάνω από 50 εκατομμύρια. Αυτό βέβαια είναι εις βάρος ανταγωνιστικότητας. Μέσα σε αυτό το τοπίο θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε περισσότερο τις υποδομές και να μην τα μεταγγελίουμε όλα στο Ναι, ναι, τελειώνω, τελειώνω, Πρόεδρε. Και παρακαλώ το Κοινοβούλιο να μελετήσει καλύτερα την πρόταση. Το ότι κάθε ρύθμιση θα πρέπει να αφορά το πώς θα ξαλαφρώσουν τα αεροδρόμια από τον κορεσμό, το οποίο θα ωφελήσει τον επιβάτη διότι θα μειωθούν τα τέλη αεροδρομίων και θα ελκύσει και από το δημόσιο και το τομέα επενδύσεις. Θα σταματήσουμε πριν τα αεροδρόμια. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Thank you. Σε ευχαριστώ. Θα δυσκολευτώ τώρα να συγκρατήσω τους βουλευτές. Γι' αυτό τουλάχιστον προσπαθώ να συγκρατήσω τους ομιλητές. Κύριε Ούγγιας, θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να κάνετε μια πρώτη παρέμβαση αν θέλετε. Ε, πέντε λεπτά μιλήστε ή τα μοιράζετε ή μια και καλή στο τέλος. Ε, εσείς ό,τι θέλετε. Πάντα. Η σημερινή συζήτηση ήταν ήδη πολύ ενδιαφέρουσα. Ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας είναι λίγος για να ακούσουμε τώρα και να πούμε όλα αυτά που δεν θέλαμε να πούμε. Γι' αυτό και είχαμε διοργανώσει και προηγούμενη ακρόαση μαζί με τη συνάδελφο που συμμετείχε και ο πρόεδρος Σίμψον και που επέτρεψε στους περισσότερους ομιλητές να έχουν περισσότερο χρόνο και να μπορέσουν να παρέμβουν. Κάναμε και μια άλλη συνάντηση με τους κοιόδης εισηγητές για να ε, μιλήσουμε ακριβώς για την... να δούμε πού βρισκόμαστε μάλλον, να κάνουμε μια επισκόπηση και νομίζω ότι μπορούμε να πούμε από αυτή την ε, φάση, ε, την διερευνητική, μπορούμε να προβούμε σε κάποιες παρατηρήσεις. Υπάρχουν ε, κάποιες, ε, κάποια σημεία από τον οποίο υπάρχει στην ουσία ελεύθερη άποψη. Υπάρχει ας πούμε η η δυνατότητα συμμετοχής όλων των πρωταγωνιστών. Υπάρχει ανάγκη διαφάνειας και ανεξαρτησίας των συντονιστών, που είναι ένα άλλο στοιχείο το οποίο αναφέρθηκε στην απόψινή συζήτηση, αλλά που ε, υπήρξε μεγάλη συνένεση από αυτή την άποψη. δευτερεύουσα τώρα αγορά των σλότ στόχο έχει να βελτιώσει την κινητικότητα των ε, χρονοθυρίδων ε, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη κινητικότητα. Γι' αυτό θεωρήσαμε ότι ήταν θετικό στοιχείο όπως και η ανεξαρτησία των συντονιστών. Καταγράφαμε λοιπόν, καταγράψαμε λοιπόν ότι ενεργούν από θέση ε, υπόλογη σε σχέση με άλλους ε, φορείς. Ε, Αφής λοιπόν διαχωρισμός λειτουργικός και οργανωτικός των συντονιστών από πλευράς των αερολιμενικών αρχών αλλά και των αεροπορικών εταιριών θα ήταν κάτι το θετικό για τη λειτουργία του συστήματος. Άλλοι τρόποι τώρα βελτιο... βελ... Ε, βελτιστοποίησης της χρήσης των ε, αερολιμενικών δυνατοτήτων και αναφέρομαι στην αύξηση του κατοφλίου χρήσης των σλότ από το 80% στο 85% και στην αύξηση της μίνιμουμ της σειράς από τις 5 ε, στις 10 εβδομάδες για τη χειμερινή περίοδο και στις 15 για τη θερινή περίοδο. Εδώ καταγράψαμε αντιπαρατηθέμενες απόψεις. Υπάρχουν συμφέροντα που έχουν δημιουργηθεί ιστορικά και που σήμερα προτάσουν διάφορα και που προέρχονται γιατί είναι ενδιαφέρον να περάσουμε από αυτή την κατάσταση. Δημιουργούνται τη στιγμή που οι εταιρείε είχαν το μονοπόλιο το πτήσεων κάθε μία εθνική εταιρεία στους ουρανούς της χώρας της ε, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τώρα πια οι εταιρείε δεν είναι εθνικές είναι ιδιωτικές και έχουμε περισσότερους ανταγωνιστές στον κόσμο της, των αεροπορικών μεταφορών. Από αυτό το σημείο αφετηρίας λοιπόν θεωρώ ότι είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε από μια κοινή θέση. Εμεί δεν, δεν έχουμε την έννοια της σλότ που θεωρείται εδώ αγαθό ε, νομικό, σε ποιους ανήκουν τα σλότ, στα έθνη, στα αεροδρόμια, στις περιφέρειες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι μια αμφιβολία την οποία πρέπει μια σχεδία παντός να τη λύσουμε. Ποια είναι η νομική θέση, φύση των σλότ. Δεν γίνεται ε, Απλώ να το αντιμετωπίζουμε ως μια διαπίστωση του τι ισχύει σήμερα και εδώ ολοκληρώνω για να μείνω στον χρόνο που μου δώσατε Πρόεδρε το σημείο για το οποίο πρέπει να μιλήσουμε. Υπόθηκε ότι από σήμερα μέχρι το 2030 θα διπλασιαστεί η κυκλοφορία των αεροπλάνων. Αν θέλουμε να, ευκαι... να εκμεταλλευτούμε αυτές τις δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης, ε, είναι ευκαιρία για θέσεις απασχόλησης, γιατί έχει προβλεφθεί μεγαλύτερη ένταξη 60.000 θέσεων απασχόλησης. Σε μια τέτοια φάση οικονομικής δυσκολίας, ε, δυσπραξίας, ε, για όλους είναι κάτι το πολύ θετικό. Αλλά θα πρέπει να γίνει με τη σωστή ισορροπία. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτήν, να μην αντιπαντήσουμε μάλλον σε αυτή την πρόκληση, γιατί αν δεν τη δώσουμε την απάντηση εμείς, θα τη δώσουν άλλοι. Είτε με την οικονομική ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και έχουμε, φέρουμε ευθύνη όλοι ε, για να δεχτούμε αυτή την πρόκληση είτε θα μας επιβληθεί από άλλους. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε για παράδειγμα ότι παντού έχουμε την απέτηση για μεγαλύτερη προστασία του περιβάλλοντος. Άρα λοιπόν η νομολογία των περιφερειακών δικαστηριών με τελευταίο αυτό της Φραγκφόρτης που <coughs> μείωσε τις πτήσεις κατά τη διάρκεια της νυχτερινής ε, περίοδου ε, είναι μια πολύ ε, ισχυρή απόφαση. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν αν θέλουμε ελεύθερη αγορά ή αν όντως τελικά θα πρέπει να περιοριστούν οι πτήσεις. Να θυμίσω κάτι ακόμα. Ο Ιταλικός κώδικας αεροπλοείας προέβλεπε το δικαίωμα επιμονής όπως ε, αποκαλείται, δηλαδή στα λιμάνια και στις παραλίες επέτρεπε σε όσους είχαν ήδη μια άδεια να μπορούν να χρησιμοποιούν, να συνεχίσουν μάλλον να χρησιμοποιούν αυτό το δικαίωμά τους. Τα εθνικά όμως δικαστήρια και το Ευρωπαϊκό Αντιτράστ επέβαλαν την κατάργηση αυτής της ρύθμισης. Ε, εάν δεν το κάνουμε εμείς λοιπόν θα μας επιβληθεί από άλλους το Κοινοβούλιο και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, όπως επαναλαμβάνω, ζητώντας και μια θεσία από την Κομισιόν, γιατί υπάρχουν υπερβολικά πολλές ε, ε, πράξεις στην πρόταση της Κομισιόν. Να αφήσουμε την μεγάλη άσκηση λοιπόν αυτών των πράξεων κατά κατεξουσιοδότηση από πλευρά της Κομισιόν θα είναι μια συμβολή σε αυτή την ισορροπία. Ευχαριστώ πολύ. Έχω τέσσερις που ζήτησαν το λόγο. Και κλείνω τον κατάλογο, άντε και ο κύριο Κοκ. Ένα λεπτό έκαστος, σοβαρά το λέω, ένα λεπτό έκαστος, κύριε Φεντάλζα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θα μείνω στην υπόδειξή σας, δεν θα σχολιάσω ούτε θα κάνω ομιλία. Θα προσπαθήσω να υποβάλω ερωτήσεις στους ε, καλεσμένους μας. Πρώτο θέμα αφορά τη σειρά των σλότ. Και ήθελα να στραφώ στον κύριο Καν πιο συγκεκριμένα. Καταλάβαμε από τη, τα slides που μας έδειξε ποιες είναι οι επιχειρησιακές δυσκολίες ε, των φορέων ενώπιον αυτού του νέου συστήματος ε, χορήγησης των ε, κατανομής των σλότ. Θα ήθελα να ανέλυε κάπως περισσότερο και το θέμα της δυσκολίας για ενδεχόμενες νέες εταιρείε που θα θέλαν να μπουν σε συγκεκριμένα σλότ. Δεδομένες της δυσκολίας να δημιουργήσει κανείς μια η αρχαιότητα, μια ιστορική παρουσία ώστε να μπορεί να ζητήσει τη συγκεκριμένη σειρά των σλότ. Κατά τη γνώμη σας λοιπόν υπάρχει μια περαιτέρω δυσκολία για τους νέους, τις νέες εταιρείες. Και η, η δεύτερη μου ερώτηση που απευθύνεται στον κύριο Φούλξ. Κυρώσεις. Εγώ πιστεύω ότι αντί να κάνουμε τα πράγματα πιο δύσκολα, θα πρέπει να ε, σκεφτούμε πιο λογικά για τις κυρώσεις. Μια υπόθεση θα μπορούσε να είναι η εφαρμογή αυτών των κυρώσεων που ορίζονται από τα κράτη-μέλη και που στόχο έχουν την ε, βελτίωση της των αερολμονικών υποδομών και όχι μόνο τον διαχειριστή τους και θα τελειώσω λέγοντας ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρόκληση που έκανε ο κύριος Μπαρόντσι για τη δευτερεύουσα εμπορία σλότς γιατί δεν θέλουμε μόνο να κάνουμε μια αγορά σλότς να βελτιώσουμε το σλότ δεν είναι η μόνη απάντηση θέλουμε και καλύτερες υποδομές και νομίζω ότι αυτή είναι μια πρόταση επί της οποίας μπορούμε και πρέπει να συζητήσουμε. Κοιτάξτε... Βοηθήστε με λίγο ρε παιδιά. Λοιπόν, ένα λεπτό, κύριε Σασόλη. Ο κύριο Σασόλη, υπάρχει, υπάρχει ένα προγραμματάκι στο iPad που λέει γίνεται Radar 24 και εκεί απευθείας μπορείτε να δείτε όλη την εναέρια κυκλοφορία αυτή τη στιγμή σε ολόκληρο τον κόσμο. Την πρώτη φορά που θα το ανοίξετε κοστίζει ένα ευρώ, πραγματικά θα σας πιάσει αγωνία. Γιατί στην Ευρώπη από πάνω γίνεται της μουρλής και αν αυτό αληθεύει ακόμη περισσότερο σε 10 χρόνια, 20 χρόνια, πρέπει να αρχίσουμε σήμερα να το σκεφτόμαστε. Αυτό το πακέτο και σημαίνει για μας, τους σοσιαλιστές δημοκράτες, ότι το κοινοβούλιο μας πρέπει να μπορέσει να το προτείνει να τα καταφέρει, γιατί είναι απαραίτητο για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. Το πρόβλημα της δευτερεύουσας αγοράς, συμφωνούμε, το θέμα των συντονιστών συμφωνούμε, καλούμε τον συντονιστή, να προχωρήσει και χρειαζόμαστε μόνο ένα πράγμα. Και κλείνω, κλείνω, μην βάρα το σφυρί, περίμενε. Μια ανάγκη έχουμε. Ευρωπαϊκούς κανόνες που να εξυπηρετούν και άλλους, κύριε να εξυπηρετούν και τους άλλους εκτός Ευρώπης. Γιατί η ενέργεια κυκλοφορία ε, συγκεντρώνεται εδώ στην Ευρώπη. Άρα και οι άλλοι θα πρέπει να λειτουργήσουν με τέτοιο τρόπο ώστε να αλλάξει η δική του συμπεριφορά. Μόνο έτσι θα έχουμε παγκόσμιες προδιαγραφές και η Ευρώπη θα έχει χρησιμεύσει σε κάτι. Ευχαριστώ. θα προσπαθήσω να τα καταφέρω. Έτσι με στυλ, έτσι, έτσι λίγο βόρειο. Όχι, όχι, εντάξει, εντάξει. Δεν θέμε να θυμώσουμε ούτε τα αεροδρόμια, ούτε να ρίξουμε τις ε, αεροπορικές εταιρείε. Μιλούσαμε για 15 εβδομάδες ε, και από την άλλη για 10. Ε, δεν μπορούμε με το 80-20 να το, να το κάνουμε κάπως όντως γιατί το 85-15 δεν βγαίνει. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Κυρία Φώστερ, για ένα λεπτάκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα είμαι τόσο σύντομη. Νομίζω πως ε, το είπαν οι άνθρωποι από το πάνελ. Χρειαζόμαστε περισσότερους ε, αεροδιαδρόμους, αλλά αυτό ξέρετε είναι σαν να λέμε πως... Ε, θα, ε, διαδρόμους προσγείωσης, με συγχωρείτε. Αλλά αυτό είναι σαν να λέμε θα σας κολλήσουμε γρήπη. Οπότε, ναι, το να παίζουμε τώρα και με τις λεπτομέρειες δεν βελτιώνει τίποτα. Δευτερογενής αγορά, την υποστηρίζω πλήρως και αν θέλω να το κάνουν και άλλα κράτη-μέλη δεν βλέπω ε, γιατί να πούμε όχι. 99% των σλότς ούτως ή άλλως αποτελούν αντικείμενο ελεύθερης εμπορίας. Οπότε μιλάμε για το 1%. Ε, επίσης, ε, το το μήκο ε, των μπλοκ, θα το αφήσω αυτό. Επίση, συντονιστέ δεν υπάρχουν σε όλα τα αεροδρόμια, αλλά υπάρχουν κάποια αεροδρόμια όπου υπάρχουν κάποια προβλήματα και εκεί πέρα πρέπει να το δούμε. Όσον αφορά λοιπόν τη λέξη κατάχρηση που ακούστηκε, Α, εντάξει, δεν είναι και τόσο εκταμένη, ίσως να υπάρχει κάποια κατάξη, εκεί πρέπει να κάνουν δουλειά οι συντονιστές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Λίχτεμπεργκερ. Θα μιλήσω Ιταλικά γιατί ίσως έτσι να μου δώσετε και ένα λεπταδάκι παραπάνω. Ναι, πάντα έτσι γίνεται. Πάντα εσείς οι ε, Ιταλοί μιλάτε δύο-τρία λεπτά. Όχι. Καλά, εντάξει, θα συνεχίσω στα γερμανικά τότε, άμα είναι έτσι. Ε, τίθεται ένα ζήτημα που ανέφερε ο κύριος Σούτζας. Σε ποιον ανήκει το σλότ. Ποιος έχει στην περίπτωση διαφωνίας την δυνατότητα να κάνει εμπορία αυτών των δικαιωμάτων. Αυτό είναι το θέμα. Βεβαίω, και αυτό είναι το ερώτημά μου προς τους τελευταίους ομιλητές, εάν υπάρχει, υπάρξει κάποια εμπορία, είναι αυτό μια λύση για το πρόβλημα, ναι ή όχι. Και αν ναι, ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτή την εμπορία, από πού προκύπτει αυτό. Ακούσαμε στην προηγούμενη ακρόαση τον Ιταλό ειδικό που ασχολήθηκε με αυτό το ζήτημα. Θέλω να παρατηρήσω, ολόκληρη η χρηματαγορά ασχολείται με χρήματα που δεν μπορεί να έχει κάποιος στην κατοχή του και δεν κατέχει. Νομικά λοιπόν, πώς το βλέπετε. Ποιο θα μπορούσε να είναι αυτός ο οποίος ε, θα μπορούσε να εμπορευτεί αυτά τα σλότ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κόχ ευτυχώς δεν θα μιλήσει, οπότε ο κύριος Γκρό μπορεί να μιλήσει για 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύντομος θα είμαι και απευθύνομαι σε αεροπορικέ εταιρείε. Εάν ε, εγώ δεν κάνω μία πτήση προς ε, το μόναχο ας πούμε και θα ε, χάσω το σλότ, τι κάνω, πετάω μισοάδιος για να διατηρήσω το σλότ ή τι ακριβώς είναι. Ευχαριστώ. Γκρός, καλά τα είπατε. Λοιπόν, κύριοι, ε, αν θέλει κάποιος να πει κάτι για δύο λεπτά, παρακαλώ. Κύριε Σμίτ, όχι, ευχαριστώ πολύ. Μόργαν, κύριε Φόξ, πού είστε, έχω χάσει την μπάλα. Δύο λεπτά. Να απαντήσω πρώτα στον κύριο Φιντάντζα. Νομίζω ότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ κύρωσης και συστήματος κράτησης των χρονοθερίδων. Λίγες είναι οι χώρες που δεν έχουν τέτοιο αποτελεσματικό, που έχουν αποτελεσματικό σύστημα όπως ας πούμε το Μήνο Βασίλειο και η Ισπανία. Και το βασικό όφελος που προκύπτει από αυτά τα δύο συστήματα είναι ότι δεν θεωρούμε ότι είναι κύρωση το σύστημα κράτηση. Είναι κίνητρο. Κίνητρο προς τις αεροπορικές εταιρείες για να επιστρέψουν έγκαιρα τις χρονοθερίδες πριν δηλαδή την ε, προθεσμία όπως προβλέπει η ΙΑΤΑ στις καθημερινές της. Επομένως, έτσι να μπορούν να ξαναδοθούν σε κάποιες εταιρείες ε, τα σλότ. Όλοι θέλουν να υπάρχει τέτοι, τέτοιου είδους προβολήτες, τέτοια, τέτοια διαφάνεια. Αν λοιπόν ε, αργά επιστρέψουν τα σλότ μία εβδομάδα πριν ας πούμε ε, από, την, από, την, ε, από την περίοδο χρήση, πρέπει να είσαι πάρα πολύ τυχερό για να το πάρει κάποιο άλλο. Ε, και επαναλαμβάνω, όχι, δε αυτό, δεν, αυτό γίνεται για να ωφεληθούν οι ευρωπαϊκέ εταιρείε. Δεν γίνεται για να βγάλουν αυτά τα αεροδρόμια. Γιατί ό,τι βγει από την επαναπόληση πάει στι εταιρείε την επόμενη, την επόμενη χρονιά. Ένα, ένα κομματάκι από τα τέλη αεροδρομίων. Ναι. Ναι, τίποτα δεν λέμε που δεν ισχύει. Ο κύριος ε, Χουσενκάν και εγώ εκπροσωπώ την Ιάτρα, ε, Ιάκα. Ε, δεν θα ανέφερα τι την Ιάτρα. Τέλος πάντων, εμείς μπορούμε να προσπαθούμε όσο μπορούμε να έχουμε διαφάνεια. Εξαρτάται, κύριε Φιντάντσα, τι ορισμό δίνει κανένα, γιατί οι περιορισμοί που αφορούν τα σλότ εδώ στην Ευρώπη, αν δείτε τι γίνεται και με το κομμάτι του κάργου στην αγορά, δείτε τι κάνουν οι εταιρείε χαμηλού κόστου κλπ. Βλέπετε τι, τι είδου πρόσβαση έχουν ή δεν έχουν. Άρα νομίζω ότι το 80-20% που ισχύει τώρα δεν εμποδίζει αναγκαστικά την πρόσβαση στην αγορά στις περισσότερες περιπτώσεις. Ίσως ε, υπάρχουν, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις που δεν μπορεί κανείς να τρυπώσει σε κάποιο αεροδρόμιο, αλλά καταρχήν δεν επηρεάζεται η αγορά με το ισχύον σύστημα. Να επανέλθουμε τώρα στον κύριο Σασόλη. Α, ναι, και οι άλλοι θα πρέπει να αλλάξουν, όντως. Ε, ε, αυτό το σύστημα έχει αποδώσει παγκοσμίω είναι αποδεκτό από όλου. Και αυτό που ε, λέω ω επιχείρημα θα πρέπει η Ευρώπη να είναι πολύ προσεκτική, μην προχωρήσει σε κάτι το οποίο έχει τοπική ισχύ και να ελπίζω ότι οι άλλοι θα ακολουθήσουν. Εγώ διατηρώ πάρα πολλέ επιφυλάξει σε σχέση με αυτό. Θα πολύ πολύ προσεκτικό. Κύριε Γκρό, αν εγώ θα πέταγα, θα, θα οδηγούσα ένα άδειο αεροπλάνο, ίσω. Αν θα το, θα, θα το δρομολογούσα. Τι να σα πω. Ναι, εγώ θα το έκανα. Δεν ξέρω αν θα το έκανα οι ευρωπαϊκέ εταιρείε. Ε, επιφυλάσσομαι για τα σλότ. Θα, είμαι πάρα πολύ προσεκτικό να αποδεχτώ πρόταση η οποία θα έδινε υπερβολικά πολλά κίνητρα. Συγγνώμη, συγγνώμη σα παντώ διπλωματικά, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μάθιος. Σας ευχαριστώ. Καλά τα πήγε μέχρι σήμερα το σύστημα και όπως ε, όλα τα πράγματα τα οποία έχουν κάνει τον κύκλο τους θα πρέπει να το δούμε ξανά και γι' αυτό και εμείς θέλουμε να δούμε σε ποια σημεία θα τροποποιήσουμε τον κανονισμό, θα τον αναβαθμίσουμε και να τον επικαιροποιήσουμε για τον 21ο αιώνα. Ε, η EasyJet έχει ωφεληθεί επομένω από αυτό το καθεστώ. συνεχίζουμε την ε, αναψητερία σε σχέση με του, του, του, του σύνων εποχή, τους νέους καιρούς και θα πρέπει να δούμε κατά πόσον ε, αν μπει πιο ψηλά ο πύχης για το νέο εισερχόμενο ε, θα είναι δύσκολο εμεί να κρατήσουμε τις χρονοθυρίδες μας αλλά εμείς για να ωφεληθούν όλοι από την βελτίωση του ανταγωνισμού είμαστε προετοιμασμένοι να αποδεχτούμε την ε, πρόκληση. Κύριε Μπαρονίτση, έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Εγώ, εγώ δεν χρειάζομαι δύο λεπτά. Απλώς θέλω να απαντήσω στην κυρία Λίχτενμπέργκερ σε αυτό που ερώτησε. Σας υπενθυμίζω ότι ETS, στην, στο, στο νομοθέτημα εκείνο, το οποίο είχατε περάσει το ETS, ήταν πολύ πρωτοπόρο και ε, από την εμπορία των εκπομπών τα έσοδα ε, ε, ήταν, προβλεπόταν να πάνε στις υποδομές. Γιατί να μην κάνουμε το ίδιο και, και όσον αφορά την εν λόγω αγορά και εν λόγω εμπορία των ε, χρονοθυρίδων δηλαδή. Θα μας πείτε τις απόψεις, ο καθένας και δική του άποψη. Έχουμε πέντε φορές απόψεις και εδώ στο πάνελ. Πάντως, για μισό λεφτάκι, με δύο λόγια. 10 εβδομάδες αντί για 50, λέει κύριε Μάισνερ δεν είναι υποχρεωτικό να γίνει έτσι. Τα εισοδήματα πάνε, τα έσοδα μάλλον, πάνε στις ε, αεροπορικές εταιρείε. Έχουν πολλά κοινά όσον αφορά αυτό οι εταιρείε και το 10 εβδομάδες αντί για 15, να το δούμε. Οι περισσότερες σειρές κρατάνε όλη τη σεζόν. Άρα να μην ε, κοιτάμε μόνο τις εξαιρέσεις. 10 παρά 15 είναι πιο λογικό ας πούμε για τη θερινή περίοδο. Σύντομα, έχετε το λόγο κύριε. Ποιο κερδίζει από αυτό το πρόγραμμα, λέει ο κύριος Έχει δίκιο ο προλαλή αλλά ο πλευρά πολιτική. εσείς, ο νομοθέτης είναι ο κύριος των χρονοθερίδων. Εσείς θεσπίζετε τους κανόνες που ρυθμίζουν το ποιο θα πάρει τις χρονοθερίδες. Εσείς έχετε λοιπόν στα χέρια σα το τιμόνι για να το χρησιμοποιήσετε καλά. Α, δηλαδή λέτε ότι ε, εμείς κονομάμε. Αυτό, αυτό θέλω να πει τέλος πάντων. Ευχαριστούμε το πρώτο πάνελ και έχουμε τώρα αλλαγές κοιτάλες. Και πάμε παρακάτω. Στις υπηρεσίες εδάφους, άλλο θέμα που και αυτό είναι επίμαχο. Πάμε τώρα στο επόμενο πάνελ. Κόλμας, Νάβας Γαρθία είναι τα μέλη αυτού του δεύτερου πάνελ. Σας υπενθυμίζω, συνάδελφοι, ότι έχουμε μία σειρά διατάξεων της πρότασης που πρέπει να συνεξετάσουμε με την Επιτροπή Απασχόλησης και αφορούν ε, την πτυχή της κοινωνικής πολιτικής γιατί αυτό είναι το, η αρμοδιότητα της ε, Επιτροπής Απασχόλησης. Πρώτα πρώτα. Έχει τον λόγο ο κύριος Δημητρή Ντεμπούρνοβιλ. Who Καθίστε εσείς δίπλα στο μοναδικό μας λάπτοπ. Are we ready to go, guys? Έτοιμοι, φύγαμε. Πάμε. Κύριε Ντεμπορνοβίλ, έχετε ένα πεντάλεπτο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δεν θα σας πω την περίληψη που είχα για τις βασικούς στόχους. Και θα επικεντρώσω την προσοχή μου σε αυτά που ρωτήσατε πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα φέρει περισσότερη αποτελεσματικότητα, θα έχουν περισσότερη ασφάλεια, καλύτερε υπηρεσίε και απαντούμε καταφατικά. Ναι, σε κάποιε τεχνικού χαρακτήρα μεταβολέ. είμαι νομικό. και να βρω το λόγο εδώ, όχι να εκπροσωπήσω κάποιον του αλλά σαν εμπειρογνώμονας. Στα μικρότερα αεροδρόμια, υπηρεσίε εδάφου ακόμα δεν διαπώνται από κάποια ρύθμιση. Εκεί δηλαδή που έχουμε λιγότερα από 2 εκατομμύρια επιβάτε και λιγότερα από 50.000 τόνου μεταφορά φορτίου. Εξαίρεση είναι η αυτοεξυπηρέτηση όσον αφορά τι υπηρεσίε εδάφου σε σχέση με τους κανόνες ενέργεια κυκλοφορία. Οπότε είναι το θέμα τώρα της επιλογής και βέβαια σε αυτά τα αεροδρόμιο έχουμε τις γενικές ε, διατάξεις δικαίου ανταγωνισμού όπως προβλέπεται τη συνθήκη. Η διαδικασία τώρα έγκρισης και οι οικονομικές συνθήκες που θα πρέπει να πληρούνται μας θυμίζουν αυτά τα οποία ισχύουν όσον αφορά την αδειοδότηση των αεροπορικών εταιριών. Και έτσι έχουμε βεβαίω κάποιο είδου ε, γραφειοκρατία, άχθο, βάρο, οικονομικό, διοικητικό, γραφειοκρατικό για του νέου ερχόμενου και βέβαια και για τι ε, ε, αρχέ. Για όλε αυτέ τι εταιρείε υπηρεσιών εδάφου και έχουμε ένα σωρό στην ε, Ευρώπη. ο περιορισμός της έγκρισης στα πέντε χρόνια ίσως είναι προβληματικός, γιατί δεν έχουμε τέτοιο, τέτοιο περιορισμό για τις αντίστοιχε υπηρεσίες των ε, ε, αεροπορικών εταιριών. Γιατί παρέχοντε υπηρεσίες εδάφους πρόκειται συνεχώς να ελέγχονται από τις αρχές. Πέραν της αδειοδότηση. Επίσης, θα έχετε παρατηρήσει ότι υπάρχει μια ανισότητα όσον αφορά την προσβασιμότητα σε σχέση με τα αεροδρόμια και αυτούς που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες. Μόνο οι τελευταίες αυτές εταιρείες ε, υπόκεινε σε κάποιους ε, περιορισμούς. Σε σχέση τώρα με τους διαγωνισμούς υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια για ε, την κατακύρωση των αδειών, ε, σε σχέση με ερχόμενους ε, που ίσως αυτά τα κριτήρια είναι ανεπαρκή σε σχέση με τους ήδη, ε, τους παλιούς στην αγορά σε σχέση με τα στοιχεία ενεργητικού, σε σχέση με τον εξοπλισμό τους και τελευταίο επίσης αλλά σημαντικό είναι η άσκηση κάποιου ενδίκου μέσου κατά των αποφάσεων που επιδικάζουν μια τέτοια έγκριση κατόπιν κάποιας διαδικασίας. Αυτό μπορεί να αναβαθμιστεί, να βελτιωθεί, να έχουμε κάποιο είδους fast track ε, ούτω ώστε να μην έχουμε φραγμούς δικαστικού νομικού χαρακτήρα. Να σας παραπέμπω στο, στο αεροδρόμιο των Βρυξελών και αυτό για λόγω κάποιων νομικίστικων ε, εμποδιών έχουμε πάγωμα. Είχαμε πάγωμα τέλος πάντων μέχρι να ε, τελεσυνδικήσει στο θέμα. Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να περιορίσει τον ανταγωνισμό και να καθορίσει αφύσικα την τιμολογική πολιτική. Τώρα χρειάζεται πιο υγιές μοντέλο ανταγωνισμού. Το δε επίπεδο ποιοτικών υπηρεσιών θα πρέπει να το σεβαστούν οι εταιρείε. Και οι εταιρείε υπηρεσιών Οπότε προσοχή μπορεί αυτό να μας οδηγήσει σε διεύρυνση της ευθύνης των εταιριών των αεροπορικών ως προς τα δικαιώματα των επιβατών. Προσοχή, να δούμε τι θέλουν και οι ασφαλιστές, μήπως ε, ουθούν στο να πληρώνουν πολύ μεγάλα ποσά. Και άρα πάμε για επαναδιαπραγμάτευση όσον αφορά τις τυποποιημένες συμφωνίες υπηρεσιών εδάφους τώρα απλώς ασφαλείας να δούμε υπόψη τι ισχύει για την ενέργεια κυκλοφορία και για την ασφάλεια όσον αφορά το λεγόμενο καθεστώς των ρυθμισμένων φορέων Θα πρέπει εδώ να δούμε πώς θα περιχαρακώσουν έννοια του μονοπωλίου. Πώς θα επίσης υπάρχει συνέχεια και συνέχιση στην παροχή των υπηρεσιών εδάφους. Λόγω με τις αεροναυτικές δραστηριότητε. Εδώ διακυβεύονται. Θα πρέπει ομένω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην οδηγεί σε κάποιο είδους έμεση επιδότηση νομικά είναι προβληματική μια τέτοια κατάληξη. Ας πούμε αυτές τις δραστηριότητες τις οποίες να αναλάβει η διαχειριστική αρχή κάποιου αεροδρομίου ή κάποιο άλλο αεροδρομίο εκτός από το ε, κάθε αεροδρόμιο το οποίο εξετάζεται. Και επίσης θα πρέπει να δούμε πώς ορίζονται οι δραστηριότητες ε, real estate, ε, αγοραπολισίας ακινήτων. κόμμα από, την, από τον αντίστοιχο φορέα της Πολωνίας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που μας καλέσατε ώστε να σας δώσουμε και εμείς ε, τη δική μας άποψη όσον αφορά τον νέο κανονισμό. Η αρχή που θα είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του κανονισμού με βάση το νομικό πλαίσιο που έχουμε στην χώρα μας έχει στόχο την καλύτερη χρήση των ε, δυνατοτήτων στην χώρα μας αλλά και στις υπόλοιπες χώρες. Καλύτερη ποιότητα δε των ε, υπηρεσιών εδάφους θα σημάνει και καλύτερη ή αυξημένες, καλύτερες ή μάλλον αυξημένες δυνατότητες στην ε, αγορά της αεροπλοείας. Το σύστημα αυτό θα σημαίνει ότι οι εταιρείε που θέλουν να μπουν στην αγορά αυτή θα πρέπει να είναι αδειοδοτημένες και ε, να ελέγχονται επί τη βάση κάποιων συγκεκριμένων κριτηρίων. Νομίζω πως τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να τα επεξεργαστούμε κάπως περισσότερο διότι υπάρχει εδώ, υπάρχουν εδώ διάφορες δυνατότητες ερμηνείας. Τώρα όσον αφορά το σύστημα της αμοιβαίας αναγνώρισης των αδειών στην Ευρώπη, το σύστημα αυτό θα πρέπει να είναι φιλικό προς τις επιχειρήσεις που θέλουν να επεκταθούν στο εξωτερικό. Στην Ευρώπη το σύστημα της αδειοδότησης θα πρέπει να το επεξεργαστούμε κάπως περισσότερο, διότι για την ώρα επικρατεί μια κάποια βεβαιότητα σε σχέση με το πώς ε, θα δίνονται, πώς θα χορηγούνται οι άδειες. εξάλλου. Υπάρχει διατύπωση που είναι καλύτερη ε, κατά τη δική μας άποψη οι δε υπεργολάβοι θα πρέπει να μπορούν να εκτελούν τις ίδιες δραστηριότητες όπως και οι κύριοι συμβασιούχοι, οι αδειοδοτημένες δηλαδή ε, εταιρείε. Όλα αυτά βέβαια σημαίνουν ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο τρόπος λειτουργίας των υπηρεσιών εδάφους, ε, καθώς και ο κίνδυνος που διατρέχουν οι εργαζόμενοι σε αυτές τις υπηρεσίες. Τα κρατημέλη θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν, για παράδειγμα, τις ε, τιμές σε περίπτωση που έχει αναπτυχθεί ε, μονοπόλιο σε κάποιο συγκεκριμένο αεροδρόμιο. Θα πρέπει να αναπτυχθούν ίσως και να επιβολούν, επιβληθούν και τέλη για τη χρήση των υποδομών. Από την άλλη πλευρά αυτό, κάτι τέτοιο θα σήμαινε περισσότερη γραφειοκρατία τόσο για τον ε, ρυθμιστή όσο και για τη ε, αεροδρόμια. Και γι' αυτό και διερωτώμεθα κατά πόσο αυτό το θέμα θα ήταν καλύτερο να το ρυθμίσουν ε, τα ενδιαφερόμενα μέρη. να μπορέσουν δηλαδή ελεύθερα να συμφωνήσουν μεταξύ τους για τους όρους και τις συνθήκες. Επίσης η Κομισιόν μίλησε για τις νεοεισερχόμενες εταιρείες. Ωστόσο, στο επίπεδο της ομάδας εργασίας, η ιδέα που παρουσιάζεται στο σχέδιο κανονισμού της Κομισιόν έγινε δεκτή. Στην ουσία σημαίνει διαχωρισμό και λήψη υπόψη των νέων εταιριών που μπορεί να ε, παρουσιαστούν. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το θέμα των ελάχιστων προδιαγραφών οι οποίες ελάχιστες προδιαγραφές θα πρέπει να θεσπιστούν εσωτερικά από τα ίδια τα ενδιαφερόμενα μέρη. Για να ολοκληρώσω λοιπόν, να πω ότι οι στόχοι που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι καλοί, είναι δικαιολογημένοι. Είδαμε μόλις πόσο πολύ θα αυξηθεί η κυκλοφορία στα επόμενα χρόνια αλλά θα πρέπει να προσέξουμε ακόμη περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο θα ε, επιδιώξουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας. Να θυμόμαστε δηλαδή ότι η γραφειοκρατία θα πρέπει να περικόπτεται και όχι να αυξάνεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Κάρλος Νόβας ε, Γκαρσία κατόπιν από την Ένωση ε, Υπηρεσιών Αεροδρομίων. Πέντε λεπτά έχετε κύριε Γκαρσία. Thank you very much for your invitation. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας. Εκπροσωπώ την ε, Ένωση Εξυπηρέτησης Αεροδρομίων που είμαστε η μεγαλύτερη ένωση ανεξαρτήτων ε, τέτοιων εταιριών δηλαδή που δεν ανήκουν σε αεροδρόμια ή εταιρείε και στόχο έχουμε να διευρύνουμε τις ευκαιρίες πρόσβασης ε, στην αγορά. Οι ανεξάρτητες εταιρείε απετέλεσαν το μεγαλύτερο παράγοντα επιτυχία τη σχετική οδηγία και σύμφωνα με την Κομισιόν είχαμε έτσι καλύτερη ποιότητα και χαμηλότερε ε, τιμέ. Κάποιε παρατηρήσει τώρα για το ιστορικό αυτή τη πρόταση. Πρώτα απ' όλα το αεροπορικό πακέτο. Διαφωνούμε με το ότι η εξυπηρέτηση εδάφου ρυθμίζεται από το ίδιο πακέτο. Είναι διακριτά θέματα και θεωρούμε πως θα πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία στο δικό μας τομέα ανεξαρτήτως των υπολείπων κλάδων, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει. Σύμφωνα με την Κομισιόν, το κόστος ε, εξυπηρέτησης εδάφους ε, είναι 5 έως 12% του κόστους των αεροπορικών εταιριών, ενώ άλλα κόστη είναι γύρω στο 6% εντός του αεροδρομίου. Αυτό σημαίνει βεβαίως πως ε, δεν θα επηρεαστεί πολύ η τιμή του εισιτηρίου. Σύμφωνα με την Κομισιόν 17% των καθυστερήσεων ε, ε, προκαλούνται από προβλήματα στο έδαφος. Αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει εξυπηρέτηση εδάφους. Τα στατιστικά του Eurocontrol δείχνουν ε, πως ε, η εξυπηρέτηση εδάφους ε, είναι υπεύθυνη για γύρω στο 5%. Τώρα, για την αυτοεξυπηρέτηση εμείς είμαστε υπέρ του περιοριστικού ε, ορισμού. Δηλαδή μια εταιρεία και οι ε, σύμμαχες εταιρείες της. Αλλιώς θα έχει μείνει πολύ μικρό ποσοστό για να μπορέσουμε να το διεκδικήσουμε και είμαστε κατά των απεριόριστων ε, δικαιωμάτων, γιατί όπως αναγνωρίζει και η Κομισιόν, ο αντίκτυπος του πλήρους ανοίγματο θα είναι περιορισμένος, οπότε δεν είναι κατανοητός αυτός ο κανόνας και οδηγεί σε αβεβαιότητα στην αγορά. Επίσης, η είσοδο στην αγορά μέσω μιας ψευδούς άδειας αυτοεξυπηρέτησης πρέπει να απαγορευτεί, όπως σκοπεύει να κάνει άλλωστε η Κομισιόν συντονιστικός ρόλος των αεροδρομίων. Έχουμε μια πολύ απλή προσέγγιση, αντιλαμβανόμαστε και δεχόμαστε τους στόχου της Κομισιόν, αλλά θεωρούμε πως πρέπει να υπάρξει διάκριση όταν δρά το αεροδρόμιο ως εξυπηρέτηση εδάφου. Ε, τότε δεν θέλουμε να μας συντονίζει ο ανταγωνιστή μα. Πρέπει να υπάρχει ένας ανεξάρτητο φορέας για αυτή τη δουλειά, Αλλιώ υπάρχει κίνδυνο για τον ανταγωνισμό. Και έτσι πλέον δεν θα ε, ισχύουν οι στόχοι του νέου κανονισμού και δεν είναι δυνατόν να ο ανταγωνιστή μας να μα επιβάλλει πρόστιμα κάθε εβδομάδα. Επίση, ο νομικός δεν επαρκεί και εδώ πέρα μα στηρίζει και η Κομισιόν. Φαίνεται όμω πω είναι εναντίον το Συμβούλιο. Κατά την άποψή μας, Ουσιαστικό είναι ο πραγματικός έλεγχο. και η έλλειψη ε, διαφάνειας καθώς και η έλλειψη επιδότησης ε, της δραστηριότητας από άλλες δραστηριότητες μπορεί να γίνεται μέσω ενός νέου συστήματος γιατί το τωρινό δεν λειτουργεί. Ο συνάδελφος, ο κύριος δικηγόρος ε, περιέγραψε την κατάσταση του ότι δεν είναι υποχρεωμένα να προσφέρουν ε, τα αεροδρόμια να υποβάλουν προσφορές ως κάτι το οποίο ε, προξενεί αντίφαση. Εμείς θεωρούμε πως είναι διακριτική μεταχείριση. Επίσης, ο αριθμός των εταιριών. Όλοι συμφωνούν πως τα αεροδρόμια πάνω από 10 εκατομμύρια επιβάτες θα πρέπει να έχουν μια τρίτη εταιρεία. Μια απέτηση αυτή, η απέτηση αυτή δεν είναι σίγουρο ότι θα ισχύσει για αεροδρόμια που εξυπηρετούν μεταξύ 5 και 10 ε, εκατομμύρια επιβάτες. Μεταθέσεις. Δεχόμαστε τις μεταθέσεις ε, προσωπικού, αλλά με δύο σημαντικούς όρους. Πρέπει να ισχύει για όλες τις εταιρείες, όχι μόνο τις ανεξάρτητες, και πρέπει να έχει τα βασικά δικαιώματα των εργαζομένων. Για να υπάρχει και η δυνατότητα βεβαίως των εταιριών να οργανώνονται. Διαφωνούμε με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή που μιλάει για ίσα δικαιώματα. Αυτό μπορεί να σημαίνει πως οι ανεξάρτητες εταιρείες θα πρέπει να αγοράζουν εισιτήρια για, τα, το προσωπικό τους που προέρχεται από αεροπορικές εταιρείες. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο προσφέρουν δωρεάν οι αεροπορικές εταιρείες. Βεβαίω, οι μηχανισμοί αυτή μετάθεσης ε, είναι ε, παράγοντας αύξησης του κόστους κανόνες τώρα υποβολής ε, προσφορών. Υποστηρίζουμε τους κανόνες της Κομισιόν για τον ρόλο της Επιτροπής Χριστών Αεροδρομίου, καθώς υπάρχει σαφής σύγκρουση συμφερόντων. Και θεωρούμε πως θα πρέπει να υπάρχει ε, διαχωρισμός των ρόλων. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Ζασάδα, έχετε την δυνατότητα να μιλήσετε για 5 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εμπειρογνώμονες για τα... τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις τους. Ή, ε, τα ανεξάρτητα συνδικάτα των υπηρεσιών εδάφους, τα ίδια τα αεροδρόμια, οι αεροπορικές εταιρείες. καθένας βλέπει από τη δική του πλευρά το θέμα. Γι' αυτό είναι και πολύ δύσκολο να συνδυάσει κανείς και να συμφιλιώσει όλες αυτές τις διαφορετικές απόψεις. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα δούμε πολύ προσεκτικά σε ένα τομέα που απασχολεί πάνω από 100.000 κόσμου. Η γενική προσέγγιση της Κομισιόν είναι νομίζω πολύ σημαντική. Αποκέντρωση, Από εμά εξαρτάται το να σχηματίσουμε το μέλλον αυτού του τομέα στην Ευρώπη. Αλλά όλα αυτά έχουν να κάνουν με το εξής. αν είχαν μεταφραστεί όλες οι προτάσεις της Κομισιόν σε κανονισμό θα είχαμε πλήρη απορρίθμιση. Η διαδικασία για την επιλογή της υπηρεσίας εδάφου και της εταιρεία που τη διαχειρίζεται είναι διαφανής. Απ' την άλλη πλευρά, απελευθέρωση θα έπρεπε να σημαίνει ελευθερία επιλογής. του καλύτερου προμηθευτή της υπηρεσίας η ελευθερία ε, παύσης της χρήσης του συγκεκριμένου φορέα. Ένα απελευθερωμένο λοιπόν τελείως σύστημα είναι δυνατόν να υπάρξει. Δεν θα σημάνει πολύ σοβαρά προβλήματα για τα ε, αεροδρόμια μας. Ας φανταστούμε ότι έχουμε την εξής πρόταση. Ελεύθερη δηλαδή διαχείριση χωρίς κανένα περιορισμό. Ένα κοινό σύστημα βασίζεται σε κοινά κριτήρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σαφής, σαφή τέλη χωρίς διακρίσεις για την πρόσβαση στην κεντρική υποδομή. Η ελευθερία επίσης επιλογής μιας εταιρείας η οποία θα χειρίζεται τις υπηρεσίες εδάφους. Ένα σύστημα σύμφωνα με το οποίο ο, διαχει... ο του αεροδρομίου θα είναι υπεύθυνο για τι υπηρεσίε εδάφου και ιδιαίτερα για τον τομέα της ασφάλειας σε περιπτώσει κρίση πάνω απ' όλα. Τέτοιο σύστημα θα ήταν ουτοπία. Όχι. Η απάντηση είναι όχι. Έτσι ε, λειτουργούν άλλες αγορές στον κόσμο. Για παράδειγμα η Ιαπωνία γιατί την χάνει να είμαι πρόεδρος της αντιπροσωπείας με την Ιαπωνία. Τι θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν, να στείλουμε το σχέδιο αυτό κειμένου πίσω στην Επιτροπή. Φαίνεται οι περισσότεροι σκιώδει αυτό να θέλουν ή μήπως θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τροποποιήσουμε το κείμενο αυτό. Εγώ θα ήμουν υπέρ της τροποποίησης του κειμένου, γιατί υπάρχουν ε, κάποιες καρλές διατάξεις και κοινέ ε, διατάξεις και στάνταρ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση των, ε, των εργαζόμενων στις υπηρεσίες εδάφους. Αυτό που θέλουμε είναι κάτι πιο φιλόδοξο όσον αφορά τον κόσμο μας. Ευχαριστώ πολύ. Οι ερωτήσεις σας τώρα, ερωτήσεις ένα λεπτό έκαστος. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Μάνα από την Επιτροπή Επασχόλησης. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι θετικό το ότι διαχωρίσαμε τις αρμοδιότητες μεταξύ της Επιτροπής σας και της δικής μας Επιτροπής, αλλά νομίζω πως τελικά θα κάνουμε κάτι από κοινού. Κύριε Γκαρσία, το ερώτημά μου. Υπήρχαν σκέψεις ε, να πούμε πως ο κανονισμός είναι πολύ βαριά ρύθμιση μπορείτε να φανταστείτε για λόγους επικουρικότητας και διαφορετικών αναγκών των αεροδρομίων να πούμε πως θα είναι μόνο οδηγία. Είναι ικανοποιητικό αυτό για εσάς. Δεύτερον, η Κομισιόν πρότεινε πως δύο μέρες επαρκούν για την εκπαίδευση του προσωπικού. Εμένα η εμπειρία μου είναι διαφορετική Ποια είναι η δική σας η απάντηση τρίτον. Ο αριθμός ε, των ανθρώπων που εξυπηρετούν τα αεροσκάφη και θα μπορούσε να ανέβει στους τρεις και ίσως παραπάνω. Έχουμε πολύ διαφορετικές εμπειρίες στα κράτη-μέλη. Τι άποψη έχετε εσείς. Σας ευχαριστώ. Ένα λεπτό ο καθένας παρακαλώ. Φλέκενστάιν. Ναι κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα λυπούμε για το ότι δεν έχουμε και κάποιον από τα ευρωπαϊκά συνδικάτα. Ε, γιατί επηρεάζονται πάρα πολύ όπως έδειξαν άλλωστε και οι εξελίξεις ε, από την άλλη. Εγώ λυπούμαι σε αντίθεση με τον κύριο Μαν για το διαχωρισμό μεταξύ των δύο επιτροπών γιατί τα ζητήματα τα οποία μπορούμε να δούμε θετικά, τα ζητήματα ποιότητας που σχετίζονται με την εκπαίδευση και κατάρτιση πλέον δεν είναι ε, αρμοδιότητά μας ως ε, Επιτροπή Μεταφορών. Τώρα γιατί τι άποψη έχω για την ιδιοκτησιακή αποσύνδεση επιπλέον εταιρείε για το αν βοηθούν θετικά τον ανταγωνισμό και τελικά τον επιβάτη. Μέχρι στιγμή δεν έχω καταλήξει, δεν το βλέπω από αυτή την ακρόαση. Μέχρι στιγμή ε, κατά πλειοψηφία ε, είμαστε πολύ επικριτικοί. Ένα σημείο όμως πρέπει να ακουστεί στη συζήτηση. Εάν πραγματικά βοηθάει τον πελάτη να το βοηθήσουμε και δεν ε, καταπιέζει περισσότερο τον εργαζόμενο. Αλλά για λόγους ιδεολογίας και μόνο δεν θα είμαστε υπέρ της περαιτέρω απορρίθμισης. Ευχαριστώ κύριος Κλίντς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Φλέκενστάιν και εγώ θεωρώ πως ε, δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε τις ε, δομές, πρέπει να τις δούμε από κοινού. Η Κομισιόν εδώ πέρα κάνει μια υπόθεση η οποία υπόθεση εργασίας η οποία είναι λανθασμένη πως όσο μεγαλύτερο το αεροδρόμιο τόσο περισσότερες εταιρείες χρειαζόμαστε να προσφέρουν υπηρεσίες δάφους. Μπορώ να σου πω, εγώ όταν πάω σε μεγάλα αεροδρόμια όπως το Heathrow ή άλλα που έχουν 8-9 εταιρείε, δεν είναι καλύτερη η εξυπηρέτηση από ό,τι αλλού. Αντίθετα, όσο πιο μεγάλο το αεροδρόμιο, τόσο πιο περίπλοκα τα πράγματα. Και αν το συνδυάσουμε και με πολλές εταιρείες ε, που προσφέρουν υπηρεσίες εδάφους, με διαφορετικές διαδικασίες, τότε είναι προβληματικά τα πράγματα. Για εμένα λοιπόν δεν υπάρχει σχέση μεταξύ του αριθμού των εταιριών ε, που προσφέρουν την υπηρεσία και την ποιότητα της υπηρεσίας αυτής. Δεύτερον, όταν κάτι πάει στραβά, πάει κάποιος στα απολεσθέντα της ε, αεροπορικής εταιρείας. Οπότε η ευθύνη ξαφνικά της ποιότητας ε, πάει στην αεροπορική εταιρεία. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Τέλος, συμφωνώ πλήρως πως εμείς πρέπει πράγματι να ε, φροντίσουμε να μην υπάρχει επιδότηση της μίας δραστηριότητας από την άλλη. Αν το κάνει π.χ. και το αεροδρόμιο πρέπει να διαχωριστούν οι δραστηριότητες. Αυτά και δεν υπάρχει χρόνος για τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Λίχτενμπεργκερ για ένα λεπτό. Ναι, επειδή ε, προφανώς στη συζήτηση αυτή μιλάτε για ιδεολογίες, να ρωτήσω. Ποια είναι η προσθέμενη αξία για τον καταναλωτή. Ποια είναι η προσθέμενη αξία για την εταιρεία του αεροδρομίου. Δεν έχει απαντηθεί αυτό μέχρι στιγμής. Γιατί το συμπέρασμα, όσο περισσότερες εταιρείε, τόσο περισσότερη ποιότητα, δεν προέκυψε από αυτά που ακούσαμε. Άλλοι παράγοντες είναι πολύ ουσιαστικότεροι εδώ πέρα. Και συμπληρωματικά. Είχαμε συζήτηση με τον Επίτροπο Κάλλα στην αρχή της ε, θητείας μας όπου υπήρχε μεγάλο, μεγάλη απορία για, τον, για την περαιτέρω απελευθέρωση. Γιατί όταν όλα τα κόμματα δεν το ήθελαν, ήταν κατά και παρόλα αυτά πάλι αυτή η πρόταση υποβάλλεται. Ευχαριστώ κυρία Φώστερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω πως ε, το έγγραφο της Κομισιόν είναι αρκετά καλό, αλλά εντάξει υπάρχει μια ανησυχία Έχουμε εξυπηρέτηση εδάφου από διαφορετικέ εταιρείε εδώ και δεκαετίε. Δεν είναι τίποτα το καινούριο. Οι μικρέ λεγόμενες λεγόμενε εταιρείε δεν το κάνουν αυτό λόγω κόστου. Γι' αυτό περάσαμε ε, στο να είναι αυτή μια ξεχωριστή δραστηριότητα. Και μετά το ερώτημα είναι τι αποφασίζουμε εμείς. Οι περισσότερες εταιρείε κοιτάνε το επιχειρηματικό τους μοντέλο και αναλόγως λαμβάνουν μια απόφαση. Οπότε είναι δύσκολο εμείς να ορίσουμε και να πούμε ανάλογα με το μέγιστο αεροδρομίου θα έχουμε τόσες εταιρείε. Εντάξει, υπάρχει ευελιξία στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου λειτουργεί αυτό. Αλλά να πω κάτι το εξή. Να σας πω πως υπάρχουν ανησυχίες όταν έχουμε τέτοιες, όταν έχουμε προβλήματα, εξαφανίζονται και ο επιβάτης δεν ε, ξέρει ποιος ε, φταίει για το πρόβλημα που έχει. Και, είναι μπαλάκι μεταξύ αεροπορικής εταιρεία και εταιρεία εξυπηρέτησης εδάφους. Αλλά όπω είπα αυτό είναι απόφαση των εταιρεών που εξετάζουν το επιχειρηματικό του μοντέλο και αναλόγω αποφασίζουν. σε ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πρέπει να ε, επιστραφεί ως απαράδεκτη η πρόταση της ε, Κομισιόν. Έχουμε συμπίεση των μισθών και εργασιακή πίεση, χειρότερες συνθήκες εργασίας, δεν ισχύουν αυτά που μας λέει η Κομισιόν όσον αφορά την ασφάλεια, χρειαζόμαστε καλύτερη κατάρτιση, ψηλότερους μισθούς και συντονισμό των διαφόρων επιχειρήσεων στο αεροδρόμιο. Γι' αυτό το κοινωνικό ζήτημα δεν είναι χωριστό από το ζήτημα των συγκοινωνιών. Ευτό ερωτώ γιατί δεν καλέσατε συνδικάτα να μας πούνε οι ίδιοι πώς έχει η κατάσταση και τι πραγματικά χρειάζονται. Ευχαριστώ. Γκάλερ, ευχαριστώ. Το ερώτημά μου προς το πάνελ. Ε, πώς έχει κάνει λάθος υποθέσεις εργασίας η Κομισιόν για το ότι 57% των καθυστερήσεων, 75% των καθυστερήσεων οφείλεται στην εξυπηρέτηση εδάφους και αυτό το οποίο μας είπε ο εκπρόσωπος Κομισιόν θε, δεν θεωρούμε πως θα υπάρξει ε, μείωση ε, των υπηρεσιών, της ποιότητας των υπηρεσιών. Δεν, θα έπρεπε να έχει κλονιστεί λίγο η πίστη σας μετά από τις τελευταίες εξελίξεις. Επίσης το ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι ε, απόψεις των εταιριών που προσφέρουν ήδη τις υπηρεσίες. Μήπως δεν τις λαμβάνουμε όντω υπόψη και μαζί με αυτούς και την πραγματικότητα. Ο κύριος Γκαρσία ε, μίλησε για ελάχιστου αριθμούς επιβατών. Εγώ σκεφτόμουν ίσως ε, τα 15 εκατομμύρια. Αυτά. Ευχαριστώ Μάισνερ. Ευχαριστώ. Δεν θα επαναλάβω τα ίδια. Θα πω ένα πράγμα. Ένα λόγο για τον οποίο υπάρχει αυτή η οδηγία. Ένας λόγος είναι παραδείγματο χάρη η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και λιγότερες καθυστερήσεις. Πείτε μας, συγκρίνεται ένα αεροδρόμιο που έχει μία εταιρεία με ένα που έχει δύο. Υπάρχουν όντως λιγότερες καθυστερήσεις, τότε ναι, να το κάνουμε. Ευχαριστώ Κοχ. Ναι, το ερώτημα απευθύνεται στον ε, κύριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είπατε Πώ τα αεροδρόμια μπορούν να ανεβάσουν τι εταιρείε σε τρει. Δεν το κατάλαβα. Μπορούν ή πρέπει. Πρέπει ε, όταν ε, δεν επαρκούν παραδείγματο χάρη τα τέλη, τι ακριβώ είναι. Ευχαριστώ κύριε Πέρκερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όλοι γνωρίζουμε πως ένας στόχος ε, των υπηρεσιών αυτών είναι να πάνε οι επιβάτες και οι αποσκευές ε, ασφαλώς από το σημείο Α και στο σημείο Β. Οπότε βασικό εδώ πέρα είναι η ασφάλεια και τα μέτρα ασφαλείας. Ποιο είναι το πλεονέκτημα λοιπόν όταν έχουμε κάποια αεροδρόμια που λειτουργούν μια χαρά με δύο εταιρείες Ποιο είναι το πλεονέκτημα που θα προσφέρουν τρει ή τέσσερι εταιρείε εξυπηρέτησης ε, εδάφου, εδάφους. Εγώ δεν το βλέπω το πλεονέκτημα. μπορείτε εσείς ίσως να με βοηθήσετε. Δεύτερον, ε, ε ακούω πως συχνά περισσότερες εταιρείε προκαλούν περισσότερα προβλήματα παρά λύνουν κάτι. Πείτε μας, ισχύει αυτό. Γιατί με στατιστικά στοιχεία αποδεικνύεται πως έχουμε περισσότερα προβλήματα με περισσότερες εταιρείε παρά με δύο. Σας ευχαριστώ Γκρός. Ευχαριστώ. Ερώτημα, δεν θέλω να παραλάβω τα υπόλοιπα. Ε, το να συνδέσουμε την απελευθέρωση με τους μισθούς θα μπορούσαμε να το έχουμε κάνει και σε άλλους τομείς, αλλά δεν έγινε δεν απελευθερώνουμε έτσι, τόσο ποτέ. Ας τα αφήσουμε αυτό στην επικουρικότητα και να πούμε πώς μπορούν να το κάνουν οι χώρες αν Οι, διαφορές, οι διαφορετικοί μισθοί λύνονται στους μισθούς που πληρώνονται. Δεν ε, λύνονται με άλλους μηχανισμούς και συγκρίνεται τα διάφορα αεροδρόμια μεταξύ τους. Επίσης ε, νομίζω πως ε, και η δική μας Επιτροπή έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και όχι μόνο η Επιτροπή Κοινωνικών ε, Υποθέσεων. Το ερώτημά μου είναι πόσο διαρκεί η βασική εκπαίδευση στην εξυπηρέτηση εδάφους. Οι δύο μέρες που αναφέρθηκαν μου φαίνονται παράλογες. Νομίζω πως χρειάζεται πέντε με 6 μήνες. Ισχύει αυτό ή κάνω λάθος. Ευχαριστώ, Λάιχτφριντ. Ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ. Δύο πράγματα. Πρώτον, εδώ πέρα η νομοθεσία αυτή παρεμβαίνει πάρα πολύ στα κοινωνικά ζητήματα, γι' αυτό θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους. Γιατί δεν καλέσατε συνδικάτα δεύτερον. Ξέρω ένα μεγάλο αεροδρόμιο, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Βρίσκεται σε μια νήσο τη βορειοδυτικής Ευρώπη Εκεί πέρα εφαρμόζονται όλα όσα έχει προτείνει η Κομισιόν και δεν λειτουργεί τίποτα. Γι' αυτό το ερώτημά μου είναι ε, πώς θα σας φανεί να απορρίψει την πρόταση αυτή το κοινοβουλίο μας. Σας ευχαριστώ κύριε Λάχιθριτ. Ε, υπάρχουν και καλύτερα, καλύτερα αεροδρόμια στο Ηνωμένο Βασίλειο από αυτό το οποίο εννοείτε εσείς. Υπάρχουν και καλύτερα. Με εντυπωσιάζει απλώ που η φήμη αυτού του αεροδρομίου είναι παγκόσμια ε, κλίμακα, παγκόσμια εμβέλεια και δεν είναι και καλύτερη. Και τώρα, δεν είστε υποχρεωμένοι να απαντήσετε, αλλά αν θέλετε κάτι να πείτε, έχετε δύο λεπτά, κύριε Μπουρδομβίλ. Ναι, ατέθη το ερώτημα ποιο θα είναι ο τελικός λογαριασμός για τους καταναλωτές και τους επιβάτες. Ποιοτικές προδιαγραφές που μπορεί να επιβάλλει η Κομισιόν στις ε, εταιρείες παροχής υπηρεσιών εδάφους θα δοθεί στους επιβάτες να μπορέσουν να ε, ε, διεκδικήσουν ε, για την καθυστέρηση ας πούμε στο χειρισμό των αποσκευών ανάμεσα στο αεροδρόμιο και την έξοδο του αεροδρομίου είναι κάτι, κάποιες άριστη, αόριστη περιοχή όσον αφορά τις νομικές δυνατότητες. Θα μπορούσε ωστόσο να συνοδευτεί από την ανάγκη από πλευρά τη Κομισιόν να ε, παρατείνει, να, μάλλον, να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για τις καθυστερήσεις ε, και του καθεξής. Ευχαριστώ. Κόμας, η κυρία Κόμας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να αναφερθώ στο θέμα του ανταγωνιστικού πλανεκτήματος, όπως αναφέρεται στο σχέδιο της ε, Κομισιόν, όσον αφορά δηλαδή την επιλογή του φορέα παροχής υπηρεσιών εδάφους. Ε, θα πρέπει ωστόσο να υπάρχουν κάποιες μήνυμα προδιαγραφές, όπως όσον αφορά την ε, ασφάλεια, αλλά και την ποιότητα ναι, ε, θα πρέπει να υπάρχει ένα ε, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα προκύψει, που θα πρέπει να μεταφραστεί σε μια καλύτερη θέση της συγκεκριμένης εταιρεία. Ο κύριος Γκαρσία. Σας ευχαριστώ. Το θέμα του αν θα είναι οδηγία ή κανονισμός είναι πολύ ε, κέρια. Τα τελευταία χρόνια είδαμε μια σταθερή ανάπτυξη υγιή ε, της αγοράς με οδηγία. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι ε, αν υπάρχουν προβλήματα εφαρμογής της οδηγίας θα πρέπει αυτά να λυθούν με άλλους τρόπους σε σχέση με την ε, κατάρτιση, πιστεύουμε ότι η βασική κατάρτιση απαιτεί δύο εβδομάδες και η επαναληπτική δύο εβδομάδες ετησίως. Και η επαναληπτική κατάρτιση συνήθως είναι εβδομαδιαία ετησίως. Τώρα, όσον αφορά τον αριθμό των χειριστών, βεβαίως εδώ οι απόψεις διαφέρουν μέσα στο ένωσή μας. Αλλά βασική άποψη είναι ότι 5 εκατομμύρια είναι ίσως ε, πολύ χαμηλός αριθμός και ίσως θα πρέπει να γίνει τοπική αξιολόγηση γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποια αεροδρόμια με 5-6 εκατομμύρια επιβάτες που είναι όμως εποχιακοί, όπου η αγορά κυριαρχείται από αεροπορικές εταιρείες οι οποίες οι ίδιες κάνουν και την ε, ε, τις υπηρεσίες, προσφέρουν και τις υπηρεσίες εδάφους. Ε, υπάρχουν επίσης κάποια αεροδρόμια όπου δεν γίνεται αδειοδότηση. Υπάρχουν, και αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχουν ορισμένα αεροδρόμια που δέχονται ή δυόμεση φορείς φορέα ή 2,5 φορείς παροχής υπηρεσιών εδάφους. Συνήθως η δυομεση φορεις παροχης υπηρεσιων άδεια δηλαδή δεν χρησιμοποιείται. Έπειτα θα είναι σαφές για όλους στον τομέα ότι θα πρέπει να υπάρχουν ε, συγκεκριμένες ποιοτικέ προδιαγραφές, πρέπει όμως να είναι πολύ ε, αυστηρές οι συμφωνίες που ήδη ισχύουν ανάμεσα στους πελάτες, δηλαδή τις αεροπορικές εταιρείες και τις ε, εταιρείες παροχής υπηρεσιών εδάφους. Γι' αυτό και θα πρέπει να προσέξουμε πολύ σε αυτό το ζήτημα. Αυτά είχα να πω νομίζω. Κύριε Μπόλτουιν, δύο λεπτά κι εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ζωντανή και χρήσιμη συζήτηση. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα-δύο σημεία. Καταρχήν θέλω να τονίσω ότι ο Επίτροπος δεν έχει υποβάλει ένα πακέτο απορρίθμισης ε, επί ιδεολογικής βάσης. Ελπίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να το ξανασυζητήσουμε αυτό. Δεν προτείνουμε την ιδιωτικοποίηση. Αυτό είναι εκτός του πεδίου της πρότασής μας και της συνθήκης. Εμείς δεν προτείνουμε πλήρες άνοιγμα της αγοράς. Προτείνουμε ένα περιορισμένο άνοιγμα της αγοράς. Και κύριε Κόχ, για να απαντήσω στην άμεση σας ερώτηση, προτείνουμε στα μεγαλύτερα αεροδρόμια αυτά που έχουν πάνω από 5 εκατομμύρια επισκέπτες, ένα περιορισμένο άνοιγμα 2-3. Μετά από τέτοιο, ε, με πολλή αξιολόγηση, εκεί έχουμε καταλήξει. Έπειτα, Λέμε ότι 75% των καθυστερήσεων οφείλονται ε, στι υπηρεσίες εδάφους. Επίσης λέμε ότι 75% ε, γίνονται και διαπιστώνονται επί τόπου του εδάφους δηλαδή και οφείλονται στις υπηρεσίες δάφους. Και κάτι ακόμα να τονίσω. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία. Να κάνουμε ένα γρήγορο γύρο του τραπεζιού για να δούμε πού κρύβεται η προστιθέμενη αξία. Για τις εταιρείε υπάρχει εδώ μεγαλύτερη επιλογή για να επιλέξουν τις υπηρεσίες εδάφους που χρειάζονται. Όχι ελεύθερη επιλογή, κάποια μεγαλύτερη επιλογή. Για τα αεροδρόμια τους δίνει την ευκαιρία να ελέγχουν κάπως καλύτερα τη χρήση των δικών τους υποδομών από τις εταιρείε, τις αεροπορικές και από τις εταιρείε παροχή υπηρεσιών εδάφου. Δεν του δίνουμε το κλειδί βέβαια για να ελέγχουν τα πάντα, αλλά κάπω καλύτερα να τα ελέγχουν. Για τι ανεξάρτητε εταιρείε παροχή υπηρεσιών εδάφου προσφέρεται μια προοπτική για θεμητό ανταγωνισμό, για ανάπτυξη και βέβαια τη δυνατότητα για να προσφέρουν θέσεις απασχόλησης για του ίδιου του εργαζόμενου και είχαμε πολλέ καλέ συζητήσει με τι ενώσει και τα συνδικάτα για αυτό το θέμα ε, πιστεύουμε πως η πρότασή μας δίνει νομική βεβαιότητα για το προσωπικό της, ε, των υπηρεσιών εδάφους σε περίπτωση αλλαγής το φορέα παροχής των υπηρεσιών αυτών. Έτσι θα επικρατούν καλύτερες συνθήκες απασχόλησης, καλύτερη κατάρτιση και μεγαλύτερη σταθερότητα στην απασχόλησή τους. Και εδώ συμφωνώ με τον κύριο Ντεμπορνβίλ ότι για τους επιβάτες υπάρχει προοπτική καλύτερης ποιότητας βελτιώνοντας τις προδιαγραφές ποιότητας ε, στο έδαφος. Κύριε Μπόλτον, σας ε, διαβεβαιώ ότι θα έρθουν τα συνδικάτα. Δεν θα ανησυχούσα εγώ γι' αυτό, επειδή σήμερα λείπουν. Κοίτα, η ερώτησή μου είναι πάντοτε πολύ σύντομη και μετά δεν την απαντάει κανεί. Υπάρχουν λιγότερε καθυστερήσει σε αεροδρόμια με μεγαλύτερη απελευθέρωση. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. αυτή είναι η ερώτηση που κερδίζει το jackpot. Το λαχείο. Εξαρτάται. Ήδη ακούσαμε την άποψη για ορισμένα αεροδρόμια στο Λονδίνο. Είναι μια άποψη την οποία συμμερίζομαι και εγώ, αλλά Μπορεί να υπάρχουν άλλοι για τα οποία θα μπορείτε να συζητήσουμε. Α πούμε, στο Μάντσεστερ είναι απελευθερωμένο το σύστημα και φαίνεται, φαίνεται να λειτουργεί καλά. Δεν μπορούμε να γενικεύουμε πάντως το, για το κατά πόσο η απελευθέρωση, η ρύθμιση λειτουργεί ή δεν λειτουργεί. Υπάρχουν αντιφάσεις και πάει ένα αεροδρόμιο. Κύριε Μπόλουιν. Εγώ ήθελα σύντομα να πω ότι η δική σας εκτίμηση είναι σωστή. Ότι δηλαδή πάει ένα αεροδρόμιο. Μπορούμε να δώσουμε παραδείγματα απελευθερωμένων αεροδρομίων που δεν λειτουργούν και τόσο σωστά και να δώσουμε και παραδείγματα μη απελευθερωμένων που λειτουργούν καλά και τούμπαλιν. Είναι αναπερίπτωση. Εμείς πιστεύουμε ότι μια μικρή αύξηση θα βοηθούσε. Με την άδειά σας κύριε Πρόεδρε, ξέχασα να απαντήσω μια ερώτηση για το αν είναι κανονισμός ή η οδηγία προτιμότερη. Ναι, σε δύο δευτερόλεπτα. Πιστεύουμε ότι ένας κανονισμός θα ήταν είναι πιο κατάλληλος εδώ, γιατί έχουμε ε, την εμπειρία αυτής της οδηγίας που βασικά απαιτεί 27 εφαρμοστικές διατάξει από 27 κρατημέλη και θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι πάντοτε πολύ ε, συμπαγές το ιστορικό της εφαρμογής. Χρειαζόμαστε καλύτερη κοινή εφαρμογή. Ευχαριστούμε πολύ. Να την παρατεί καλή συζήτηση για τις μεταφορές και τώρα πρέπει να προχωρήσουμε στο θέμα του θορύβου. Και πάλι λοιπόν θα αλλάξετε θέσεις μεταξύ σας. Our experts this panel Και έχουμε τώρα τον κύριο Άνταμ από την Ένωση Ευρωπαϊκών Αερογραμμών, την Καστέλ Νταμάρα από την, το, τοφορέ για των αεροδρομίων, τον Μάρτιν Κέσελ, Ευρωπαϊκή Ένωση κατά των ε, παρενοχλήσεων που έρχονται από τα αεροπλάνα. If you could sit. We have, we have three and there's enough places. Yeah, but it, it stops them. If they've not got a presentation, it stops them. They can sit over there.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 Ο πρώτος από τους εμπειρογνώμονές μας είναι ο κύριος Άνταμ, την Ένωση Ευρωπαϊκών Αερογραμμών. Έχετε πέντε λεπτά, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνετε, ούτως ώστε να μπορέσει να ακουστεί η φωνή των Ευρωπαϊκών Αερογραμμών επί της προτάσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να συζητήσουμε το κείμενο αυτό από πλευράς της διεθνής πολιτικής και ξεκινούμε με τις επιφυλάξεις που ε, διατηρούμε πριν σας πούμε τις ε, προτάσεις μας. Τώρα, όσον αφορά της εναέρια, την αέρια κυκλοφορία, η ΚΕΟ το, το, έχει χτενίσει το κείμενο, ε, που είναι η φορέας του ΟΗΕ που ασχολείται με, την, με τις μεταφορές και ξεκινήσαμε το 1944 και έχουμε ως αρμοδιότητα την κανονικότητα, αποτελεσματικότητα, ασφάλεια ε, των πτήσεων αλλά και τα θέματα σχετικά με το περιβάλλον. Και κάποιες ε, χώρες ε, δέχτηκαν να μα δώσουν μόνο τέτοιε νομοθετικέ αρμοδιότητε γιατί θεωρούν ότι αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να υπάρχει ομοιογένεια και αυτό επίσης είναι μια, μια, μια, μια εγγύηση. Οπότε αυτές τα διεθνή πρότυπα δεν αρκούν τόσο ώστε να μπορούμε να έχουμε την, το επίπεδο εναρμόνιση που θέλουμε. Χρειάζονται επίση κάποια πιστοποιητικά, ή κάποιε άδειε και θα πρέπει αυτά να αναγνωριζόνται παντού. Και ο Γάλλος πιλότος του θα πρέπει να μπορεί να πετάξει στην Κίνα και ο Αμερικανός ξέρω εγώ στη Γερμανία. Αλλιώς οι διεθνείς αερομεταφορές δεν θα ήταν δυνατόν να γίνουν, τουλάχιστον όχι με το επίπεδο ασφαλείας που το οποίο απολαύουμε σήμερα και γι' αυτό και θέλουμε ε, να, να αντιταχθούμε σε οποιοδήποτε μέτρο το οποίο βαθμία θα καταργήσει κάτι το οποίο γνωρίζεται από όλου. Γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν ε, τελείω αντίθετο με τι αρχέ τη ε, ΚΕΟ. Και αυτό υπονομεύει και τις εταιρείε και σαμποτάρει τη διεθνή συνεργασία για τι ενέργειες μεταφορέ. Πάντως υπάρχουν κάποια άλλα ε, κάποιες άλλες διατάξεις που προτείνονται και ε, έτσι θα, έχουμε, θα εναρμονιστούμε, θα δυναμιστούμε με ό,τι που διεθνώς προβλέπεται όσον αφορά ας πούμε τη διαχείριση του παράγοντα θόρυβος. Ε, κάποιο σημείο της πρότασης υποχρεώνει τις τοπικές αρχές να έχουν ενιαία διαδικασία λήψης αποφάσεων και επομένως πάσα εναλλακτική εξερα, εξετάζεται και όλες οι επιπτώσεις μελετώνται και όλοι οι μπλεκόμενοι πρέπει να συνοηθούν. Και αυτό έχει σχέση με τη διερήνη του Εθνούς Δικαίου που δίνει εξουσία στην Επιτροπή να δει κατά πόσο οι τοπικές αρχές ετήρησαν ότι έπρεπε. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυτό το δικαίωμα επομένω ελέγχου και όταν το 2010 έκανε τη σχετική συμφωνία με τη ΣΥΠΑ. Και ζητείτε ότι οι αρμόδιες αρχές πρέπει να διαβουλευτούν με όλους εμπλεκομένους. Οπότε έτσι η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα βοηθήσει στο θέμα του περιορισμού του, του από το, το θόρυβο. Όμως θα πρέπει να μην ε, υπάρξει ανάμειξη με το έργο των τοπικών αρχών ε, και θα πρέπει να μην υπάρχει αυθαιρεσία, θα πρέπει ε, να μην βάλουμε ως πρώτη προτεραιότητα τον οικονομικό παράγοντα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλες τις μεταβλητές και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να έχουμε λιγότερο περιορισμό. Ε, στόχος του κανονισμού όμως δεν είναι αυτό. Δεν θέλουμε ούτε να αυξήσουμε ούτε να μειώσουμε αυτό τον περιορισμό. Οι επιδόσεις μας σε σχέση με το περιβάλλον δεν έχουν να κάνουν με ε, την ποσότητα των ε, των, των περιορισμών για να μπορέσουμε αυτές οι επιπτώσεις να, να, συγκρατηθούν θα πρέπει να δούμε όλες τις λύσεις και να μην λάβουμε υπόψη μόνο τον περιορισμό που θα περιορίσει την κινητικότητα. Οι ευρωπαϊκές αερογραμμές επομένως ζητούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ε, βοηθήσουν τόσο ώστε να είναι ορθολογική αντιμετώπιση ε, της διαχείρισης του θορύβου στα αεροδρόμια. Όμως ε, έχει κάποιες διεθνείς δεσμεύσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση και αν θεωρούμε ότι δεν αρκούν να τα αλλάξουμε, αλλά δεν μπορούμε να, ε, μην τηρήσουμε τα συμπεφωνημένα και να, να, διαφορήσουμε για αυτά που έχουμε συμφωνήσει. Δεν είναι τώρα η κυρία Κριστέλ Νταμάρ. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ κύριοι βουλευτές ε, και εμείς θα πρέπει να σας πούμε τι, τι, τι πρεσβεύουν τα μέλη της, του φορέα μας και προσαγωγικά θα πρέπει να σας πω ότι τα μέλη μας καταλαβαίνουν πάρα πολύ βαθιά το τι επιπτώσεις υπάρχουν από τις δραστηριότητες των αεροδρομίων γιατί επί πολλές δεκαετίες αυτό είναι το θέμα μας, με αυτό ασχολούμεθα και τα μέλη μας ε, ασχολούνται με όλα αυτά γιατί θεωρούμε ότι το κρόπνο συμφέρον μας είναι ε, να καλυφθούν οι ανησυχίες σχετικές του, του κόσμου. Ε, ο συνάδελφος που έλαβε το λόγο προηγουμένως σας είπε κάποια πράγματα αλλά εγώ θα σας πω ποιες είναι οι συνέπειες για τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Πρώτα πρώτα, τι θα πει η ισορροπημένη προσέγγιση. Γνωρίζουμε ήδη τις τέσσερις μεταβλητές προγραμματισμός, μείωση θορύβου και περιορισμός όσον αφορά την λειτουργία. Πρώτη για μια διαδικασία η οποία επιτρέπει στην αρμόδια αρχή να λάβει σήμερα μια απόφαση και να μπορεί και αύριο όμως να λειτουργεί το αεροδρόμιο. Πολύ σημαντικό αυτό. Ένα άλλο στοιχείο για αυτή την ισορροπημένη προσέγγιση, ότι είναι η μόνη διαδικασία που μας βοηθά να μειώσουμε το θόρυβο χωρίς να προεξοφλείται με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό. Επίσης, απόφαση που θα ληφθεί θα ληφθεί υπόψη στη μελέτη των επιπτώσεων αλλά μπορεί να μην εφαρμοστεί. Um, in order to illustrate the importance of the balanced approach, I would like to focus... Τώρα, με τη σειρά μου. Να σας πω... Όπου οι τοπικές αρχές θεωρεί ότι είναι στατική σημασία στο τοπικό αεροδρόμιο, θα πρέπει να λάβει ό,τι πιο πρόσφορο μέτρο υπάρχει σε σχέση με τι δραστηριότητε του αεροδρομίου και τους τριγύρω κατοίκους. Να, στην Βαλονία υπήρχε στρατηγική άποψη για το αεροδρόμιο της. Και ρύθμισα ανάλογα τις νυχτερινές πτήσεις. 500 εκατομμύρια ευρώ ξόδεψαν για τη διαχείριση της υπαίθρου γύρω Ανανέωση του στόλου. είναι κάτι το οποίο βοηθάται όταν έχουμε τέτοιου επενδύσει. Αντίστοιχα ρυθμίζεται και το θέμα του θορύβου. Στο χήθρο, α πούμε. Άλλο παράδειγμα. Ο αριθμό, των κατοικιών εκεί αυξήθηκε 7% μεταξύ 1991 και 2009 γιατί έγινε καλή χωροταξική πολιτική και πολιτική σχετικά με την ανοικοδόμηση των ακινήτων. Επομένω υπήρχε μια ισόρροπη προσέγγιση, σωστά εφαρμόστηκε. Επομένω το θέμα είναι κατά πόσο μπορεί να έχουν σωστό προγραμματισμό οι αρμόδιε αρχέ. Τώρα, ποια είναι η προσθεμένη αξία που προκύπτει από την πρόταση της Κομισιόν. Μα αρέσει. μα δίνει τη δυνατότητα να έχουμε ισόρροπη προσέγγιση, όπω είπε και ο Μισελ, αλλά αλλά ταυτόχρονα διαχειρίζονται το θέμα του, του θορύβου αλλά και του αεροδρόμου γενικά οι αρχές διαχείρισης του αεροδρομίου. Και έχουμε μέσα τους εξής διάβλους να λύσουμε το πρόβλημα. Πρώτα-πρώτα, νομοθεσία. Αν υπάρχει ενιαία διαδικασία στην Ένωση, αυτό γίνεται με κάποιον κανονισμό. Αλλά επίσης υπάρχει το άρθρο 10, το δικαίωμα ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να σας πω δύο λόγια σε σχέση με αυτό. μπορεί η Κομισιόν να, ε, να προσφύγει στην διαδικασία επί παραβάση, αλλά αυτό δεν βοηθάει για τα αεροδρόμια. Γιατί αν ξεκινήσει διαδικασία επί παραβάση η Κομισιόν, αυτό θα γίνει αφού έχουν περιορισμό τη λειτουργία του αεροδρομίου και εάν διώξει κανείς μια αεροπορική επιχείρηση αυτή δεν γυρίζει ποτέ πίσω. Ούτε επίσης μπορεί να πει στον κόσμο. Περιορίσαμε την αεροδρομία και τώρα θα την ξαναρχίσουμε. Άρα, πάρα πολύ σημαντικό το άρθρο 10. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να εξετάσει κάποιο μέτρο πριν αυτό εφαρμοστεί. Για το θόρυβο. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η επικουρικότητα. Πρώτον, γιατί η αξιολόγηση του θορύβου γίνεται από τις αρχές του αεροδρομίου. Δεύτερον, είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει πρόβλημα, το το υπάρχει δεν υπάρχει πρόβλημα, με το θόρυβο θα πρέπει να το στις αρχές επίσης. Και πάλι όσον αφορά το περιβάλλον και το θόρυβο θα πρέπει οι τοπικές αρχές να αποφασίζουν. Το άρθρο 10 είναι πάρα πολύ σημαντικό, το χρειαζόμαστε γιατί αυτό θα μας οδηγήσει σε μια πραγματικά εξισορροπημένη προσέγγιση και δεν θα έχουμε μια ντεκαφεϊνέ εκδοχή της όπως ήδη συμβεί, αποδυναμωμένη, απονευρωμένη. Σας ευχαριστούμε Δευτέρη και τώρα. Επόμενο, επόμενος είναι ο Μαρτίν Ρέσελ από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του θεωρίου Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πρώτη φορά που οι άνθρωποι οι οποίοι ενοχλούνται από το θόρυβο μπορούν να μιλήσουν ενώπιον του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής σας. Ευχαριστώ για την ε, πρόσκλησή σας. Είναι ευκαιρία να εξηγήσουμε τις απόψεις μας. Η οργάνωσή μου είναι παλαιότατη Ε, ιδρύθηκε από τους ε, προκατόχους μας ε, το 1968 ήδη όταν δεν σκεφτόταν κανείς την προστασία του περιβάλλοντος. Είμαστε μοναδικός, η μοναδική ευρωπαϊκή μικιό. Δεν υπάρχει λόμπι για το θέμα μας. Έχουμε μέλη σε 8 χώρες και 30 ευρωπαϊκά αεροδρόμια και είμαστε μέλος άλλων οργανώσεων και χαιρόμαστε για το ότι μπορούμε να να λάβουμε μέρος στη διαδικασία στην ομάδα εργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Αεροδρομίων. Γιατί εκεί πέρα εξετάζεται το τι χρειάζεται ως δυναμικότητα αεροδρομίων. Γιατί υπάρχει αυτό, παραδείγματος χάρη για τους αυτοκινητόδρομους, αλλά όχι για τα αεροδρόμια και ακόμα και στα κράτη-μέλη έχουμε καταστάσεις άγριας δύση. Από εδώ και από εκεί ξεφυτρώνουν, κλείνουν αεροδρόμια και δεν υπάρχει εθνική πολιτική. Θα να αναφερθώ σε τέσσερα ζητήματα. Έχουμε την περιβαλλοντική ικανότητα ενός αεροδρομίου, τη φέρουσα αν θέλετε ικανότητα, ποια, ε, ποιο είναι η επέκταση μπορεί να έχει ένα αεροδρόμιο και αυτό το οποίο η ΚΑΟ λέει λεγόμενη ισορροπημένη προσέγγιση. Ο στόχος μας ως ε, οργάνωση ανθρώπων που ενοχλούνται είναι πως θέλουμε μακροπρόθεσμο σχεδιασμό των αεροδρομίων στην Ευρώπη. Αυτό δεν υπάρχει. Και η συνέπεια είναι πως από εδώ και από εκεί υπάρχουν δυνατότητες όπως λέγονται και σε κάποια σημεία έχουμε προβλήματα Would be more planning, but there is no planning. που θα λύνονταν βεβαίως με κάποιον σχεδιασμό. Δείτε παραδείγματος χάρη την Κολονία, το Χίθρο, το Παρίσι αν ε, υπήρχε σχεδιασμός ε, για το κάργο τη νύχτα δεν θα είχαμε πρόβλημα. Αν πήγαινε κάποια κίνηση, κάποιες πτήσεις δηλαδή, ε, σε άλλα μέρη που δεν ζουν άνθρωποι από κάτω. Η δυνατότητα λοιπόν, η ικανότητα η περιβαλλοντική είναι είναι και οικονομικό ζήτημα αν μπορεί δηλαδή ένα αεροδρόμιο να αναπτυχθεί, αλλά η ικανότητα αυτή πρέπει να αναπτυχθεί μαζί με τους πολίτες που ζουν γύρω-γύρω και ενοχλούνται από το θόρυβο. Και έχουν το πιο αρνητικό... Αυτός είναι ο πιο αρνητικός αντίκτυπος αυτή τη στιγμή της αεροπορίας. Στόχος μας είναι να μειωθεί ο θόρυβος των αεροσκαφών και αυτό θα το επιτύχουμε με περιορισμούς. Η λεγόμενη ισορροπημένη προσέγγιση του ΙΚΑΟ δεν είναι ισορροπημένη κατά την άποψή μας. θα μπορούσε να είναι ισορροπημένη εάν όσοι ενοχλούνται από το θόρυβο και δεν μπορούν να κοιμηθούν γέροι, νέοι, παιδιά, πάνω από 10 εκατομμύρια άνθρωποι που ενοχλούνται, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να κοιμηθούν τα βράδια, αν ε, γίνονταν σεβαστοί και έβρισκαν μια ισορροπία. Αλλά δεν το βλέπουμε. Είμαστε σε μειονεκτική θέση οι περιορισμοί στη λειτουργία έχουν βεβαίως το αμεσότερο και καλύτερο αποτέλεσμα. Ξέρουμε πως υπάρχουν διάφοροι τρόποι μέτρησης, αλλά ο αποτελεσματικότερος είναι να γίνει κάτι με περιορισμούς, όπως στη Φραγκφούρτη παραδείγματος χάρη, όπου μπορούμε να κοιμηθούμε από τις 11 μέχρι τις 5 το πρωί. Εγώ όλη μου τη ζωή Ζω 5 μίλια από τα αεροδρόμια τη Φραγκφούρτη. Ε, Επιτέλου μπορώ να ξανανοίξω το παράθυρο. Και αυτό είναι μεγάλο πλέον για κάποιον που ζει δίπλα σε ένα αεροδρόμιο. Και ελπίζουμε και αλλού να συμβεί το ίδιο. Έχουμε 240 αεροδρόμια στην Ευρώπη. Αλλά το πρόβλημα είναι στο 10% που δεν υπάρχει ρύθμιση. Ε, μπορεί να ρυθμιστεί, αλλά όχι με την αυτή προσέγγιση της Κομισιόν που συζητάμε σήμερα. Επίσης, τι άλλο δεν υπάρχει στο αεροπορικό αυτό πακέτο. Δεν ε, είναι σύμφωνοι οι περιορισμοί με αυτά τα οποία έχει θέσει η ίδια η Κομισιόν για ε, το θόρυβο και ο στόχος μας είναι οι άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται τοπικά να διαπραγματευτούν κάποιους συμβιβασμούς με τα αεροδρόμια να έχουν τοπικούς περιορισμούς για τις τοπικές ανάγκες που διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Αν δούμε 240 αεροδρόμια στην Ευρώπη, ε, ένα αεροδρόμιο στη Βόρεια Φιλανδία διαφέρει από ε, ένα αεροδρόμιο της Μαγιόρκας, ας πούμε, ή της Βαρκελόνης ή το Λινάτε στην Ιταλία ή τα μεγάλα, ξέρω εγώ, τα, τα πέντε μεγάλα σε Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία και Ολλανδία αν φροντίσουμε αυτές τις ανάγκες και έχει ο κόσμος τη δυνατότητα να το ρυθμίσει ή να συνεχίσουν οι ρυθμίσεις που υφίστανται. Γιατί υπάρχουν ήδη τοπικοί κανόνες, τότε έχουμε τη δυνατότητα στο μέλλον να έχουμε μία μείωση του θορύβου. Σημαντικό για εμάς είναι το ότι οι πολίτες της Ένωσης πρέπει να έχουν προτεραιότητα σε σχέση με τους οικονομικούς στόχους ε, των εταιριών. Η πρόταση που έχουμε τώρα, τι στόχο έχει. Πρώτα απ' όλα την ανάπτυξη του αεροδρομίου και δευτερεύον ε, ζήτημα είναι η μείωση του θορύβου και η δυνατότητα κάποιων να ξανακοιμηθούν. Ε, δεν είναι σωστό αυτό. Εμείς θέλουμε να αναθεωρηθεί το σχέδιο και οι κανόνες περί να βασιστούν στις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και να απαγορευτούν οι νυχτερινές πτήσεις για 8 ώρες σε όλα τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank Εμείς ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα ο επόμενος του μας, ο τελευταίο είναι ο κ. για 5 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε πριν ξεκινήσω να κάνω μια παρατήρηση για αυτά τα οποία ο κύριος Κέσλερ. Δύο παρατηρήσεις. Πρώτη, είναι αυτονόητο πως και οι άνθρωποι οι οποίοι επιβαρύνονται ή ενοχλούνται από το θόρυβο να, είναι στις ακροάσεις. Αλλά γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελείται μόνο από βιομηχανίες αλλά και από τα συμφέροντα των πολιτών. Και έτσι είναι τα πράγματα αυτό το οποίο όμως θα ήθελα να πω είναι πως οπωσδήποτε ε, έχετε την θέση σας εδώ πέρα, ψηφίζετε ευρωβουλευτές και οι ευρωβουλευτές σας εκπροσωπούν εδώ πέρα. Τώρα, όσον αφορά την πρόταση της ε, Κομισιόν, συνολικά να αναφέρω τρία πράγματα. Εγώ υπέρ της χρήσης της ισορροπημένης προσέγγισης επί της αρχής. Δεν την έχουμε συζητήσει αρκετά. Επίσης θεωρώ πως πρέπει να γίνει μια λογική επανεξέταση υπό όρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θεωρώ πως πρέπει να το συζητήσουμε και εδώ πέρα υποστηρίζω την ομοθετική πρόταση αυτή, αλλά θα μπορούσε χρόνο να μειωθούν τα αεροσκάφη ε, τα οποία εκπληρώνουν τις προδιαγραφές της κατηγορίας 4. Αλλά ήδη σε αυτή την πρόταση βεβαίως ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες και πρέπει να τη συζητήσουμε σοβαρά. Αν συζητήσουμε τώρα την προσέγγιση που έχουμε εδώ πέρα, έχουμε πάλι το εξής φαινόμενο. η Κομισιόν δεν είναι ουδέτερη όταν λέει ισορροπημένη προσέγγιση οπωσδήποτε και ο ανταγωνισμός και τα οικονομικά συμφέροντα λαμβάνονται υπόψη, αλλά αναφέρει από την άλλη και το ζήτημα της υγείας, της προστασίας των γειτόνων. Αλλά μας λέει μετά πως έχει οριακή οικονομική σημασία. Ε, όχι, δεν πάει έτσι. Πρέπει να είναι ουδέτερη η Κομισιόν να μην υπάρξει αυτή η στάθμιση που κάνει των δύο αντικρουόμενων αυτών συμφερόντων. Τώρα για το ζήτημα της ε, επανεξέτασης ε, νομοθετημάτων στο τοπικό επίπεδο, εάν θεωρητικά ισχύει. Μα εδώ πέρα δεν έχουμε μια καθαρά νομοθετική διαδικασία ε, Έχουμε μία μακροσκελή διαδικασία λήψη αποφάσεων με συμμετοχή των πολιτών, πρωτοβουλειών, πολιτών. που εκτείνεται σε έτη ολόκληρα και στο τέλος αυτής της διαδικασίας καταλήγουμε σε ένα αποτέλεσμα όπου όλοι οι συμμετέχοντες είναι ως ένα βαθμό ε, ικανοποιημένη. Τι θα συνέβαινε λοιπόν εάν η Κομισιόν ε, μπορούσε να ξανανοίξει αυτές τις διαδικασίες σύμφωνα με το άρθρο 10. Δεν θα βοηθούσε αυτό στη δημοτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οπωσδήποτε και στο τέλος. Όταν γίνεται μια διαδικασία που διαρκεί χρόνια και κάπως ικανοποιούνται όλοι, ποιο το νόημα μετά να ξανανοίγει η υπόθεση και να γίνουν τα πάντα διαφορετικά πρέπει να σκεφτούμε τι είναι πραγματικά λογικό. Εκεί δε που δεν συμφωνώ καθόλου και θα σας το πω ξεκάθαρα και δεν αντιλαμβάνομαι την πρόταση της Κομισιόν είναι τα ουσιαστικά μέτρα για το μέλλον που επηρεάζουν την ποιότητα της ε, νομοθεσίας ε, και δεν μπορεί αυτά να τα ξεπετάμε ως ε, πράξεις κατεξιοδότηση. Όταν στο μέλλον θα ε, ορίζουμε τα όρια θορύβου, αν θα εγκρίνονται ή δεν θα εγκρίνονται τύποι αεροσκαφών. Εγώ θα ήθελα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να το κάνει ως νομοθέτης και να μην είναι ε, η αρμοδιότητα αυτή της πράξης κατ' Σας το λέω ξεκάθαρα, δεν βλέπω δηλαδή τη λογική εδώ πέρα. Σύνοψίζοντας θα έλεγα, ε, η πρόταση της ε, Κομισιόν δεν πετυχαίνει το στόχο. Πρέπει να αλλάξει, να την αλλάξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με πολλή δουλειά θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάτι το λογικό. Αλλά δεν θα είναι απλά τα πράγματα και πρέπει να σου το πω ξεκάθαρα με τις πολλές πολλές συζητήσεις που έχω κάνει με τους συναδέλφους έχω την αίσθηση πως ούτε αυτή η εύκολη αντιμετώπιση της ε, Κομισιόν βοήθησε στην επικριτική διάθεση πολλών συναδέλφων. Δεν θα ήταν ε, αναγκαίο όλο αυτό το οποίο. Θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε ένα λογικό αποτέλεσμα, αλλά δεν είμαι σίγουρος εάν θα επιτύχουμε. Σας ευχαριστώ. Κύριο Μαν από την Επιτροπή Απασχόλησης. Θα ήθελα να υπενθυμίσω πως εμείς πάντα λέγαμε πως χρειαζόμαστε ρύθμιση από τα δικαστήρια για το θόρυβο. Ξέρετε κύριε Κέσελ πως αυτό συμβαίνει στη Γερμανία και όπως είπε και ο κύριος έχετε την δυνατότητα και δικαίως να έρχεστε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί λέμε ε, όταν έχουμε επιτύχει συνενετικά απαγόρευση των νυχτερινών πτήσεων πρέπει να τηρείται κιόλας. Και να ακούγονται και οι γείτονε πράγματι κύριε Λάχη αλλά να πω πολλοί από μας ε, ξέρετε και εγώ μιλήσαμε με πρωτοβουλίες πολιτών τα παίρνουμε πάρα πολύ σοβαρά αυτά τα πράγματα και είναι ουσιαστικό κριτήριο. Τώρα, αεροπορική κίνηση των αεροδρομίων. Κοιτάξτε, ε, η προτεραιότητα είναι η αγορά ή... Η αγορά επομένως ε, και από την άλλη μεριά είναι οι άνθρωποι, να δούμε επομένως, δηλαδή ποιες είναι οι πιθανότητες που υπάρχουν ούτως ώστε ε, να συνδυαστεί ε, ε το μεν συμφέρον με το δε. Και επομένω πρόκειται για κάποιες αλλαγέ. Και έτσι να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά την ασφάλεια και γι' αυτό θέλουμε ε, να, είναι και, να υπάρχει κάτι που συμφωνηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να είναι αποκρισταλωμένο και να μην έχουμε κάθε τρεις και λίγο κάποιες αλλαγές, διότι αυτό δημιουργεί ε, ανασφάλεια στον κόσμο. Ευχαριστούμε κύριε Γκάλερα, έχετε ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ ε, εγώ Πρόεδρε και θα ήθελα να σας πω ότι για την περίπτωση του θορύβου από θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι να κάτσουν γύρω από το τραπέζι και να βρουν ε, ε, κάποια γλώσσα συνεννόησης και έτσι να προκύψει κάποια λύση. Το θέμα είναι τι γίνεται εάν η συνένεση που θα διαμορφωθεί δεν αντιστοιχεί στην λεγόμενη ισορροπημένη προσέγγιση. Ποιος θα κρίνει, ποιος θα κατησχίσει. Εγώ, πιστεύω ότι θα πρέπει να απαλληφθεί το άρθρο 10 σε σχέση με το κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να κρατεί τα ενία σε αυτή τη διαδικασία ανάλογα με το τι θέλουμε να πετύχουμε κάθε φορά ε, στη γειτονιά ούτως υπήν του κάθε αεροδρομίου. Μήπω θα μπορούσαμε να πετύχουμε μόνο στο ίδιο αποτέλεσμα με άλλα μέσα. Δηλαδή, να αναθεωρηθεί η υπάρχουσα οδηγία ή ο κανονισμός να λάβει υπόψη τις συγκεκριμένες συνθήκες του κάθε τόπου. Ο επόμενος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα εγώ θα ήθελα να μάθω το κόστος. Ποιο θα είναι αυτού του κανονισμού, δηλαδή τι θα, τι, θα κοστίζει το να απογραφούν οι χτερινές πτήσεις. Κανείς δεν είπε τίποτα γι' αυτό μέχρι τώρα. Μήπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να, να μας πει ποιες θα είναι οι επιπτώσεις από αυτές της πλευράς. ποιο θα είναι το κόστος ε, για όλους και τους μη Ευρωπαίους, τις μη ευρωπαϊκές ε, Λύσεις δεν υπάρχουν, ούτε και για το θέμα του θορύβου στην Ευρώπη. Χρειάζεται μια ισόρροπη αντιμετώπιση, γιατί έτσι οι τοπικές αρχές θα πρέπει να έχουν εναλλακτικέ. Να μην έχουν σαν μόνη, μόνη καταφυγή τους περιορισμούς των πτήσεων. Η χρήση της γης, η διαχείριση κλπ. Τέλος, είμαι φεντρελιστής και είμαι υπέρ του δικαιώματος ελέγχου. Γι' αυτό και η εξισορροπημένη αντιμετώπιση θα πρέπει να οδηγήσει στα μέτρα που είναι τα πιο πρόσφορα, τα αυτά που φέρνουν καλύτερη σχέση κόστο αποτέλεσμα και μην πάμε αναγκαστικά στι απογραφέ των πτήσεων. Κοίτα, θεωρητικά όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι εκτεθειμένοι, είναι ευάλωτοι στη, στην, στα αυθαίρετη λύση. Τέλο πάντων, θεωρώ ότι έχει θετικό πνεύμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ω προ τα συμμετών των εμπλεκομένων. Λίχτενμπεργκερ, ευχαριστώ. Ισορροπημένη προσέγγιση. Η προσέγγιση δεν είναι ισορροπημένη γιατί εκ των προτέρων ε, ε, είναι σημαντικότερη η οικονομική παραγωγή. Μετά μας λέτε χωροταξία. Τι να κάνουμε όταν έχει ληφθεί μια λανθασμένη απόφαση στο παρελθόν. Όλοι οι γείτονε ε, που είναι εκατοντάδε χιλιάδε θα την πληρώσουν γιατί έγινε ένα λάθο στο παρελθόν. Ε, δεν είναι δυνατόν. Ε, λάθο. Είναι λάθο σκεπτικό. Τα μέτρα τα οποία προτείνονται μετά. Τι είναι εκεί πέρα κάτι πασαλήματα. Το έχω παρακολουθήσει ίδια σε πολλές περιπτώσεις επόμενο ζήτημα ε, επικουρικότητα. Αυτό γίνεται με πολλές δυσκολίες, επιδιαιτησίες και τα λοιπά και βρίσκεται μια δύσκολη λύση μεταξύ αεροδρομίου και γειτόνων. Γιατί για το όνομα του Θεού μετά από όλη αυτή τη διαδικασία έρχεται η Κομισιόν και λέει όχι απαγορεύεται. Ε, δεν είναι αρκετά δύσκολη διαδικασία. Το απορρίπτω λοιπόν αυτό. Και τελευταία ερώτηση. Το παράδειγμα το οποίο αναφέρατε για τη Βαλονία. Ε, δηλαδή, εάν η επιλογή είναι ε, να επενδύσουμε 500 εκατομμύρια και μετά να σκεφτούμε ε, επένδυση στην προστασία από το θόρυβο, δεν είναι, δεν είναι λογικό αυτό. Και ποιος είναι υπεύθυνο δηλαδή για αυτό το πράγμα. Κυρία Φώστερ, ευχαριστώ. Θα συμφωνήσω με τον Μάικλ Γκάλερ για τις πράξεις κάτι εξουσιοδότηση και το ζήτημα αυτό του ότι ήταν κανονισμός και τώρα έγινε οδηγία. Υπάρχει ζήτημα επικουρικότητας και παρά το ότι υπάρχουν προβλήματα από καιρούς καιρών πρέπει να παραμείνει η τοπική ε, συνεισφορά. Συμφωνώ προφανώς με την ισορροπημένη προσέγγιση, πρέπει να συμμορφωθούμε με τις διεθνείς προδιαγραφές. Ανησυχώ για το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αποφασίζει πως αυτή πρέπει να αποφασίσει τι είναι το οριακά συμμορφούμενο. Δεν είναι δουλειά της. Το να πάμε από τα 10 στα 5 δεσιμπέλ θα προσγειώσει στόλους ε, αεροσκαφών ε, όπως τα α380 και τα 747 πράγματα παράλογα. Επίσης αν δούμε ελαφρυντικούς ε, παράγοντες, ε, λίγα σχόλια γίνονται για τον Σεζάρ, ε, την τεχνολογία που αναπτύσσεται, τους καθαρούς ουρανούς, αυτά τα οποία κάνουμε εδώ και δεκαετίες. Κοιτάξτε, εγώ όταν μετακόμισα τέσσερα μίλια από το Χίθρο ήξερα πως υπήρχε ένα αεροδρόμιο δίπλα μου και δεν είναι τα πράγματα σήμερα όπως ήταν πριν από 35 χρόνια, σας βεβαιώ. Πρέπει αυτά και αυτές οι συζητήσεις να γίνονται σε εθνικό επίπεδο. Σας ευχαριστώ. Ε, κυρία Μελής, για ένα λεπτό. Ναι, κοιτάξτε, εγώ θεωρώ πως η υγεία πρέπει να έχει προβάδισμα έναντι των οικονομικών συμφερόντων. Ξέρω πόσο δύσκολη είναι η απαγόρευση των νυχτερινών πτήσεων να επιτευχθεί δηλαδή και δεν είναι δυνατόν η Κομισιόν να τα ανατρέπει όλα. Στο Αμβούργο, στην πόλη μου, ε, υπάρχει αεροδρόμιο της ε, πόλης που επηρεάζει πάρα πολλούς ανθρώπους και ή στη Φραγκφούρτη, εκεί πέρα επηρεάζεται ολόκληρη η περιοχή Μάιν, Ρήνου, στο Δε, Βερολίνο, ξεσηκώνονται οι κάτοικοι κατά του νέου αεροδρομίου. Για τον κανονισμό διαχείρισης ε, ε, θορύβου μας λέτε πως ε, είναι δουλειά των κρατών μελών. Και η Γαλλική Γερουσία και η Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή είναι κατά. Πρέπει να μειωθεί ο θόρυβος των ε, αεροδρομίων. Συμφωνώ με τον κύριο Κέσελ εδώ πέρα. 8 ώρες ε, νυχτερινή απαγόρευση. Ή δεν ξέρω, η Κομισιόν τι θέλει να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι να κοιμούνται με κλειστά παράθυρα. Κύριε Γκρός. Καλά. Τώρα τι να πω για τη Βαλονία υπέρ ή κατά. Ε, δώσαμε 25.000 ε, ευρώ ανακάτοικο για να φτιάξουμε ένα αεροδρόμιο που δίνει 6.000 δουλειές. Μπορούμε νομίζω να γεφυρώσουμε την οικολογία, την οικονομία και την ευτυχία των κατοίκων των γειτόνων. Έχουμε ησυχία στο αεροδρόμιο της Λιαγής γιατί όλες αυτές οι συνεννοήσεις έγιναν από πριν και για μένα αποτελεί κορυφαίο παράδειγμα στην Ευρώπη, στην Ευρώπη επένδυσης. wissen, da Να σας πω, ακριβώς αυτό το παράδειγμα, γιατί εκεί πέρα επικρατεί η ειρήνη, η η πρόταση αυτή λοιπόν δεν μπορεί να διαταράσει την ειρήνη που επιτεύχθηκε μετά από πολλές συζητήσεις και ε, διαιτησίες. Αυτός είναι ο φόβος των ανθρώπων. Δεν είναι δυνατόν. Θέλω εδώ πέρα σαφή απάντηση από την Κομισιόν. Μάλιστα τέλος. Κουν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Θα τηρήσω το ένα λεπτό. Τα κράτη-μέλη έχουν νόμους περιορισμού για τις εκπομπές και τις εκπομπές θορύβου και για δισιμπέλ ε, και απόσταση από τα σπίτια και ε, εκεί πέρα πρέπει να παραπέμπει και αυτός ο οργανισμός δεν μπορεί να ανοίξει δυνατότητα να υπάρξουν παραθυράκια και βέβαιως πολλές κινήσεις πολιτών έχουν, ε, είναι κατά των ε, πτήσεων, ε, αλλά ναι, μπορούμε και να καταργήσουμε τελείως τις και πράγματι έτσι θα έχει επιτευχθεί ο στόχος κατάργησης της ενόχλησης. Αλλά κοιτάξτε, στη Ζηρίχη παραδείγματο χάρη, μέτρησαν ακριβώς, έβαλαν κάμερες στο διάδρομο προσγείωσης, σε κάθε προσγείωση και απογείωση. Και το μεταδίδουν στα σπίτια το μεταδίδουν στα σπίτια για να βλέπουν ε, ποια είναι η ένταση του θορύβου. Γιατί καμιά φορά είναι και υποκειμενικό. Για να μπορούν, καταλαβαίνετε τι σας λέω, μεταδίδουν τα δεδομένα σε ζωντανό χρόνο για να τα ξέρουν οι γείτονε ότι τηρείται ο νόμος. Έτσι, διαφάνεια και έλεγχο και συμπεριλάβετε τους πολίτες. Σα ευχαριστώ τώρα η δική μα για δύο λεπτά ο καθένα αν θέλετε να απαντήσετε κύριε Ραντάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να απαντήσω σε τρία, τρεις παρατηρήσεις που έγιναν. Η πρώτη αφορά το ότι υπόθηκε πως οι οικονομικές, ε, οικονομικοί προβληματισμοί και οι προβληματισμοί κερδοφορίας είναι αυτοί που υπερισχύουν κάθε φορά. Στο κείμενο δεν λέει πουθενά ότι το πιο αποτελεσματικό από τους ε, κείμενο είναι αυτό το οποίο προτιμάτε. Είναι πολύ διαφορετικά αυτά τα στοιχεία και αν δούμε ε, την ισορροπημένη προσέγγιση έχουμε, θα δείτε ότι έχουμε διαφορετικούς ε, ορισμούς. Βλέπουμε το κόστος κάθε μέτρου μας επιτρέπει την επίτευξη του στόχου. Cost-benefit είναι κάτι διαφορετικό. Έχει μόνο το στόχο υπό το φω του κόστου. Και εδώ το κείμενο είναι σαφές. Μιλάει για κόστος-οφέλεια. Ε, ζητείται δηλαδή οικονομική αποτίμηση και τίποτα παραπάνω. Έχουμε τοπικά παραδείγματα, ε, προσωπικές εμπειρίες, η κατάσταση είναι διαφορετική. Γιατί λοιπόν να μιλάμε για μια λύση η οποία στην ουσία είναι η απαγόρευση νυχτερινών πτήσεων 8, ε, 8 αυτή είναι μια απόφαση που πρέπει να ληφθεί από τις τοπικές αρχές. Ο στόχος δεν είναι να υποκαταστήσουμε εμείς τις ε, τοπικές αρχές και τις αποφάσεις τους. Θέλουμε μόνο να πλαισιώσουμε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Και τέλος, επανερχόμενοι, σε αυτά τα τοπικά, στα τοπικά παραδείγματα, θέλω να ολοκληρώσω, αν δεν τον πειράζει το Πρόεδρο, με ένα προσωπικό παράδειγμα. Εγώ ζω σε, πάνω σε μια λοφόρο, πολύ σύχναστη. Φυσικά και με ενοχλεί ο θόρυβος της κυκλοφορίας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα ζητήσω να κλείσουν οι δρόμοι στην κυκλοφορία σε όλες τις Βρυξέλλες. Υπάρχουν άλλες λύσεις. Ίσως θα μπορούσαμε να δούμε τα παράθυρα, την απομόνωση των ε, παραθύρων ε, ή να δούμε τα πεζοδρόμια που απορροφούν τον ήχο, την ηχορύπανση. Μπορούσαμε να βρούμε λοιπόν λύσεις για όλα τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Κυρία Νταμάρα, δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τούμας μου απίθυνε μια ερώτηση. Αλλαγή των αεροδιαδρόμων. Και για το κανδυνός προς το χήθρο θέλουμε να κάνουμε μια καινούργια χωροταξία για να ρυθμίσουμε την ευξημένη κυκλοφορία. Κάποιες λύσεις για να μειώσουμε τις επιπτώσεις της κυκλοφορίας γύρω στα αεροδρόμια. Με νέο αεροδιάδρομο ίσως αντί για τους προηγουμένους να ενοχλήσουμε άλλους, αλλά θα είναι λιγότεροι. προηγήθηκε ο Ευρωπαϊκός Ουρανός και η εφαρμογή του που είχε κάποιες συνέπειες. Επομένως, ό,τι μεταβολή θα, θα, θα κάνουμε θα αποσκοπεί στο να ενοχλούνται λιγότεροι. Και ό,τι και αν φασίσουμε θα προηγηθούν διαβουλεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους πολίτες. Αυτούς που ενοχλούνται από το θόρυβο. Τώρα όσον αφορά το κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να παρίσταται την εκφραστική αρμοδιότητα στη, στη διαδικασία συνένεση. Έχω να σας δώσω παράδειγμα την Βιέννη, που είναι παράδειγμα προς μίμηση για την διαβούλευση που κρατά εδώ και μία δεκαετία. Δεν υπάρχει κανένα φόβο για το αεροδρόμιο που να προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα, η διαδικασία θα έχει σημασία και όχι μόνο το αποτέλεσμα. Και επομένως όλα αυτά πιστεύουμε ότι θα οδηγήσουν σε ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Κύριε Κεσίλ, ένα δίλεπτο παρακαλώ, λέει ο Πρόεδρος. Όχι, όχι δεν δίνω το λόγο. Απλώ, συμφωνεί δεν συμφωνεί. σε, σε παρακαλώ να μην γκρινιάζει. Κύριε Κέσσελ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ για τι ερωτήσει σα. Η βασική διαφορά μεταξύ του θερικού από το τρένο ή από το αεροδρόμιο ή από το δρόμο είναι ότι δεν μπορεί να αποφύγει το το αεροδρόμιο. Αν κανένας αγοράσει σπίτι πάει να μείνει δίπλα σε γραμμές, σε δρόμο, ξέρει τι θα έχει. Αλλά κανείς δεν ξέρει ποια μέρα ο αεροδρόμος θα πέρασει πάνω από το κεφάλι του. Δηλαδή κανείς επενδύει σε ένα ακίνητο, αλλά ενδεχομένω. Εκεί που δεν υπήρχε πρόβλημα σήμερα θα υπάρξει αύριο. Δηλαδή δεν μπορούμε, δεν μπορείτε να, να, τον, να τον αποφύγετε όποτε συμβεί αυτό. Δεύτερον, οι αρνητικές συνέπειες του θορύβου από τα αεροπλάνα έχουν οδηγήσει σε υψηλές δαπάνες για την κοινωνία και για της ασφάλειας. Είναι δεδομένο ότι αυτός ο θόρυβος προκαλεί υπέρταση για και άλλες ασθένειες. Άρα και αυτό θα πρέπει να το λάβει υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν θέλει να προχωρήσει προς τη θέσπιση του σχετικού κανονισμού. Εμείς προτιμούμε οδηγία και όχι κανονισμό. Κύριε Μπόλγουιν, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Και αυτή η συζήτηση πολύ χρήσιμη. Και ε, άκουσα τι είπατε. Κύριε Λέχτιν. Μάλλον ο κύριος Λάχφριντ. Θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε τις ανησυχίες σας. Τώρα όσον αφορά τα αεροπλάνα. Δεν μπορούμε εμείς να αποφασίσουμε. σχέση με αεροπλάνο θα κάνει λιγότερο θόρυβο. Προσπαθούμε να ακολουθήσουμε τα πρότυπα της ε, ΑΕΚΟ. Να βρούμε μια λύση είναι καλή σχέση κόστο αποτελέσματο και να θεσπίσουμε μια πολιτική, ένα μέτρο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα αεροδρόμια εάν καταλήξουν ει περιορισμού πτήσεων. Και θέλουμε να είναι κοινοί οι κανόνε που να μπορούν να χρησιμοποιήσουν αεροδρόμιο εάν οδηγηθεί σε περιορισμό των πτήσεων. Τώρα, οι συγκεκριμένε ειδικότερε συνέπειε εξαρτώνται από το ποιο αεροδρόμιο θα διαλέξει αυτό το, αυτή τη λύση. το, άλλο το οποίο συζητήθηκε, το κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποφασίσει για τον εαυτό της τον ρόλο του, να έχει τον ρόλο του χωροφύλακα. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Ε, μετά, ποιος θα επικρατήσει όταν έχουμε αντιφατικά, συγκρουόμενα συμφέροντα. Σαν το Σολομόντο λοιπόν θα αποφασίσει αν προσφύγουν αυτοί στην ε, Κομισιόν. Όχι βέβαια. Εμείς απλώς θα ελέγχουμε το εάν έγιναν όσα τάση, ως προϋποθέσεις η, οδηγία. Όχι, όχι, όχι, ο κανονισμός διορθώνει. Έγινε διαβούλευση. Συμμετέχω στη διαβούλευση ιδέοντε. ιδέοντες. Άλλοι είπαν ποια είναι η πιο σωστή προσέγγιση προς κόστος αποτελέσματο. Δεν είναι ο ρόλο μας αυτός. Εμείς θα, το, το, δηλαδή Επιτόπου αποφασίζεται το αν, είναι, αν ε- λήφθησαν υπόψη τα αντιφατικά συμφέροντα. Εάν οι ντόπιοι που δεν μας νοιάζει να είναι να είναι αποδοτική η λύση, είναι δική τους, δικό τους θέμα. Δεν αποφασίζουμε εμείς από αυτού. Άρα ο καθένας θα πρέπει να αποφασίσει και οι ντόπιοι θα αποφασίζουν επίσης για λογαριασμό τους. Και η διαδικασία θα είναι εκείνη η οποία προβλέπεται. Αυτή που θα συμφωνήσουμε. Το θέμα είναι τώρα, αν χρειαζόμαστε κανονισμό ή ε, οδηγία, ό,τι και να κάνουμε, θα θέλουμε να καταλήξουμε σε μια ρύθμιση κοινή για όλου. Κύριε Μπόδικο, να ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο και τώρα να ευχαριστήσω όχι μόνο του τρει εμπειρογνώμονε του τελευταίου πάνελ, αλλά όλου όλους του ειδικού που ήρθαν και μας μίλησαν ε, σήμερα. Να ευχαριστήσουμε επίσης τους βουλευτές οι οποίοι συμμορφώθηκαν με τα χρονικά όρια των αγορεύσεων, ήσαν λακωνικοί, εδώ τελείωσε η ακρόαση. Ευχαριστούμε και τους εισηγητές και τους κοιόδης εισηγητές. Δεν έχουμε τίποτε άλλο. Σήμερα τη μεσία διάταξη. Επομένως, το μόνο που μένει να σας πω είναι το που θα συνδυάσουμε την επόμενη φορά. Στις Βρυξέλλες. Δευτέρα 30 Μαΐου. 3 η ώρα. Ευχαριστούμε και τους ε, διερμηνείς. Ευχαριστούμε και τους κλητήρες, του Σουισχέ. Γιατί, Γιατί πάνε μπρος πίσω, γύρω γύρω, όταν αλλάζουν ε, οι ομιλούντες, αλλάζουν ε, τα καρτελάκια. Οπότε εκτός από τους διερμηνείς να ευχαριστήσουμε και τους κλητήρες. Κλείσω το πέρα της συνεδριάσεως.